Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καθίστε σας παρακαλώ. Σας άφησα λίγα λεπτά, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε αν θέλουμε να τελειώσουμε και στην ώρα μας. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην ακρόασή μας αυτή όσον αφορά την παράκτεια και μικρής κλίμακας αλία. Όπως γνωρίζετε όλοι, εν ώψη της ε, μεταρρύθμισης της κοινή αλλιευτικής πολιτικής, η Επιτροπή Αλίας μας αποφάσισε να οργανώσει διάφορες δημόσιες ακροάσεις για το κάθε θέμα που τόσο πολύ ενδιαφέρουν την Επιτροπή μας. Ένα από αυτά είναι η παράκτεια και μικρής κλίμακας αλίας και θέλουμε να ξέρουμε τι ρόλο μπορούμε να παίξουμε στη μεταρρύθμιση αυτή προκειμένου να βελτιώσουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δεξιάγεται η αλή αυτή. Πάνω από 80% τα νούμερα είναι ξεκάθαρα των σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτω των 12 μέτρων. Προς το παρόν αυτό είναι το όριο για να θεωρηθεί μια αλία μικρής κλίμακας. Επίσης οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της αλίας αυτής είναι τεράστιες για πάρα πολλές περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εξαρτώνται από την αλία. Και υπάρχει και κάτι άλλο που θέλω να υπογραμμίσω εδώ και είναι ότι δεν υπάρχει κεφαλοποίηση όσον αφορά την ε, αλία στα νυχτά. Οπότε χρειάζεται εδώ ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά και την χρηματοδότηση αλλά και την διαχείρισή της. Νομίζω ότι είναι σημαντικό λοιπόν σήμερα να σας ακούσουμε, να συζητήσουμε μαζί σας και να μάθουμε από σας κυρίως από τους προσκεκλημένους μας λοιπόν που θέλουμε να απαντήσουν στις ερωτήσεις που όλοι θέτουμε. Καλώς ορίσατε. Ελπίζω η ακρόαση αυτή, όπως είπα, να αποδειχθεί πολύ χρήσιμη για το έργο της Επιτροπής μας. Θέλω λοιπόν ευθύ αμέσω να δώσω το λόγο σε όσους παρουσίασαν την μελέτη που τους ανέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα χαρακτηριστικά αυτού του είδους αλία, δηλαδή η παράκτια και μικρής κλίμακας αλίας. Είναι ο κύριος Μακφάιντεν και ο κύριος Σάλς. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο ή αν και οι δύο θα πάρουν το λόγο. Πάντως καλώς ήρθατε και σας παρακαλώ. Ε, ξεκινήστε για να μας παρουσιάσετε το θέμα, όχι πάνω από 20 λεπτά όμως, γιατί αλλιώ μας πιέζει ο χρόνος και θέλουμε να ακούσουμε και τους προσκεκλημένους μας, τους άλλους. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Thank you very much for the... Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την ευκαιρία που μου προσφέρετε να παρουσιάσω αυτή τη μελέτη σήμερα και πριν αρχίσω θα ήθελα να σα παρουσιαστώ. Το όνομα μου είναι Γκρέ Μακφάντιν και είμαι πρόεδρος, διευθυντής του Ποσειδώνα που είναι μια εταιρεία, Poseidon μάλλον, που είναι μια εταιρεία η οποία μελετά και την ευρωπαϊκή αλλά και την διεθνή αλληλεία και ο Πάβελ Σάλτ από την εταιρεία Framian που είναι εταιρεία συμβούλων, ειδικά για τα θέματα της αλληλείας. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε σήμερα το απόγευμα είναι να παρουσιάσουμε τα κέρια σημεία αυτή τη μελέτη που μα ανατέθηκε εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και που ολοκληρώθηκε το πρώτο εξάμεινο αυτού του έτου. Η μελέτη αυτή ε, έδωσε, βασίστηκε στην ε, παραγωγή και στον όγκο της Ευρωπαϊκής Αλλίας και έδωσε το ένασμα διαφόρων αντιδράσεων οι οποίες άπτονται της ε, κοινή αλληλευτικής πολιτικής και των διαφόρων πτυχών και προβλημάτων. Έχουμε λοιπόν Δύο είναι οι βασικοί συμπράκτες ε, σε αυτή τη ε, μελέτη. Εγώ θα κάνω την εισαγωγή και μετά ο Πάβελ θα σας, ε, θα σας εξηγήσει τη μεθοδολογία και οι δυο μας θα κάνουμε μια σύντομη ανασκόπηση της αλλιές μικράς κλίμακας και ο Πάβελ θα κάνει και μια ανάλυση των συγκεκριμένων ε, ε, συγκεκριμένων τόπων της, της και, ε, και οι δυο μας πάλι θα σας παρουσιάσουμε ό,τι τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στις περιοχές ΝΑΤΣ 2 και τον περιφερειακό ρόλο αυτών των δεδομένων και θα παρουσιάσουμε και τα συμπεράσματα. Η μελέτη μας δεν είχε στόχο να να ξεκινήσει μία ολόκληρη συζήτηση αλλά να επικεντρωθεί ε, στις, στην παραγωγή, στον όγκο της αλίας και να παρουσιάσει στοιχεία που θα χρησιμεύσει γενικά στη συζήτηση. Η στόχη λοιπόν της μελέτης αυτής ε, ήταν να παρουσιάσει μία ενισχυμένη κατανόηση της φύσης ε, των αλλιευτικών στόλων μικρής κλίμακας, για την αλία μικρής κλίμακας Αναφερθήκαμε ειδικά στο, στα χαρακτηριστικά των αλλιευτικών δραστηριοτήτων, την οικονομική απόδοση και το ρόλο των ε, αλλιευτικών στόλων για την αλλία μικρής κλίμακος στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός, αυτός ήταν ο στόχος, η εντολή που μας ανατέθηκε. Χωρίσαμε τη μελέτη μας σε δύο τμήματα. Ο πρώτος, ε, ε, το πρώτο μέρος αναφερόταν στην τυπολογία του αλλιευτικού στόλου βάσει του επίπεδου NATS 2 και στα χαρακτηριστικά του, των στολίσκων βάσει των ε, αρχείων των ε, καταχωρήσεων του των ελευτικών στολίσκων στα αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, εξετάσαμε τους στολίσκους, τα υλικά, την ηλικία τους κλπ. Ο, το δεύτερο τμήμα της μελέτης εξετάζει σε περισσότερες λεπτομέρειες την οικονομική απόδοση και τον ρόλο της αλίας μικρής μικρής κλίμακας και γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε και τα αρχεία των στολίσκων αλλά και τα στοιχεία που υπάρχουν μέσα στην οδηγία πλαίσιο και στοιχεία της Eurostat για την απασχόληση και την ανεργία και τα εισοδήματα. Ίσως ε, προσέξετε την προηγούμενη διαφάνεια που αναφερόταν στο στόχο αυτής της μελέτης, ε, προσπαθήσαμε να επεκτείνουμε λίγο το περιεχόμενο της μελέτης εκτός του πεδίου αναφοράς, του, του πεδίου ισχύω που μας είχε δηλαδή δοθεί, για να δώσουμε τη δυνατότητα ευρύτερη ανάλυσης των στοιχείων μας. Δίνω τώρα το λόγο στον Πάβελ για να μας προσιάσει μερικά από τα αποτελέσματα. Σε ευχαριστώ, Γκραμ. Η μελέτη βασίζεται σε τρεις πηγές ε, δεδομένων. Το αρχείο του αλλιευτικού στόλου της κοινότητας, όπου χρησιμοποίησαμε πληροφορίες που ήταν κατοχωρημένες στο, περίπου στο στο μέσο του 2010, οπότε είναι σχετικά πρόσφατα και ενημερωμένα τα στοιχεία μας για την αλία μικρής κλίμακος. Δεύτερον, τα οικονομικά στοιχεία που προέρχονται κυρίως ε, από την εφαρμογή του κανονισμού ρύθμισης των δεδομένων ε, και περιέχουν κυρίως οικονομικά στοιχεία, κόστος, εισόδημα, εισοδήματα, αριθμός αλλιών κλπ. Ε, και για την Eurostat, η οποία μας ε, παρουσίασε, μας έδωσε στοιχεία για την παραγωγή και τα εισοδήματα της περιοχής ΝΑΤΣ 2. Επικεντρωθήκαμε κυρίως στην αλία μικρής κλίμακος και χρησιμοποιήσαμε και τα στοιχεία μιας άλλης μελέτης που είχε γίνει πριν απο δυο 2-3 χρόνια. Κάναμε χρησιμοποίησαμε επίσης και τη μελέτη επιπτώσεων η οποία παρουσιάστηκε όταν ε, έγιναν οι τελευταίες προτάσεις για την κοινή αλλιευτική πολιτική και διάφορες άλλες ε, πηγές όπως ας πούμε ε, εταιρείες, σύνδεσμοι, ενώσεις αλλιέων κλπ. Ε, χρησιμοποίησαμε επίσης ε, πυρογνώμενε ε, και συμβούλους από άλλες χώρες. Δεν είναι δυνατόν να συλλεχθούν όλα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, αλλά βασικά μας ενδιαφέρει η μικρή αλία, η αλία μικρής κλίμακας της περιφέρειας ΝΑΤΣ 2. Έτσι, μπορέσαμε να μελετήσουμε την σχετική κατανομή των στόλων, των ελευτικών στόλων σε αυτή την περιφέρεια. Διότι τα στοιχεία που βασίζονται ή προέρχονται από τον κανονισμό ε, των δεδομένων δεν καλύπτουν συγκεκριμένα την περιφέρεια ΝΑΤΣ 2. Όσον αφορά τώρα τα αρχεία, Καταχώρηση του στόλου χρησιμοποίησαμε, έκαναμε μία ανάλυση δύο βασμίδων SSP2 ε, και χρησιμοποιήσαμε διάφορες μαθηματικές τεχνητές, τεχνικές ε, τις οποίες ευτυχώς δεν χρειάζεται να σας αναλύσω γιατί υπάρχουν ε, στάνταρ λογισμικά τα οποία χρησιμοποιούνται η αλία μικρής κλίμακα στην Ευρώπη, εδώ βλέπετε ακριβώς τι αντιπροσωπεύει. Κατά τα μέσα του περσινού, του περσινού έτους, περίπου 83% ε, των, των ελευτικών στόλων, στολίσκων κλπ. Ε, εκτελούσε αλία μικράς, μικρής κλίμακας. Ενώ σκάφη κάτω από τα 12 μέτρα. Η, ο στόλος μικρής ε, κλίμακας ε, αντιπροσωπεύει το 10% του ε, τονάζ, του γενικού τονάζ του αλευτικού στόλου. Τα τελευταία 10 χρόνια τα σκάφη της αλίας μικράς κλίμακας μειώνονται σταθερά και έχουν μειωθεί κατά 20% την τελευταία δεκαετία περίπου 70.000 σκάφη περίπου 20% μείωση λοιπόν του στόλου μικρής κλίμακας. Η πιο σημαντική στόλη για αλληλεία μικρής κλίμακας είναι στην Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Γαλλία. Και αυτές οι πέντε χώρες καλύπτουν το 67% του συνόλου του στόλου αλληλείας μικρής κλίμακας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, τα, ο μέσος όρος των χαρακτηριστικών ε, αυτού του στόλου είναι 5-7 ε, μέτρα μήκο τα σκάφη, ε, τονάζ 3, ε, 3 τόνοι κατά μέσο όρο και ε, ε, ισχύς μηχανής 34 κιλό βατ, 34 και χρησιμοποιούν κυ, κυρίως uh, only 10... ζήκτια και παραγάδια. πελαγικές πελαγικές, είναι πελαγικές μηχανότρατες κυρίως. Ε, στο χάρτη αυτό βλέπετε τη γενική κατανομή των ε, στόλων μικρής κλίμακος ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς οι μαύρες περιοχές είναι οι περιοχές με τα μεγαλύτερα, μεγαλύτερο αριθμό σκαφών και βλέπετε ότι αυτό το κατόφλι ε, παρουσιάζεται στις Βαλτικές χώρες, στη Βόρειο, στο Βόρειο Ενωμένο Βασίλειο της Σκοτία, Ιρλανδία και βεβαίως στην Βυρική Χερσόνησο και τέλος στην Ιταλία, Σικελία, Σαρδινία και το, το, το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδος. Εδώ έχουμε και στη Βουλγαρία. Ε, εδώ έχουμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση λοιπόν μικρού στόλου, μικρής κλίμακας αλίας. Ε, περιοχές παράκτιες είναι βεβαίως αυτές. 22 από αυτές τις παράκτιες περιοχές έχουν, ε, τέσσερις έχουν πάνω από χίλια σκάφη και πολύ λίγες παράκτιες περιοχές έχουν ε, τη, τη μικρότερη συγκέντρωση σκαφών. Αυτή η πυκνή, η πυκνή συγκέντρωση ε, ε, ε, σκαφών μικρής αλίας, μικρής κλίμακας δεν σημαίνει ότι η αλία μικρής κλίμακας είναι και εξαιρετικά παραγωγική σε σχέση με τις περιοχές όπου υπάρχει λιγότερη πυκνότητα του στόλου αυτού. Μας ζητήθηκε να σχεδιάσουμε μια τυπολογία του αλλιευτικού αυτού στόλου ανάλογα με τις περιοχές συγκέντρωσης, με αυτά τα clusters. Καταρχάς λοιπόν έχουμε εντοπίσει 400 περιφερειακά ε, κλάστερς, 400 περιφερειακές τέτοιες τοπικές συγκεντρώσεις ε, σκαφών και χρησιμοποιήσαμε συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης. Ε, τα, τα τρία αυτά κριτήρια είναι ο βασικός εξοπλισμός, το μήκος και το υλικό κατασκευής των σκαφών. Επιλέξαμε αυτά τα κριτήρια διότι συνδέονται βασικά με τα άλλα τέσσερα κριτήρια τα οποία έχουμε χρησιμοποιήσει ε, για την αξιολόγηση της μεγάλης αλίας ή της πελαγικής αλίας. Ο, το μήκος του σκάφους έχει απόλυτη σχέση με τη δύναμη, την ισχύ της μηχανής και την κατασκευή του ε, υλικού, του εξωτερικού υλικού και σημειώσαμε ότι τα παλαιότερα σκάφη είναι κυρίως ξύλινα. 6 με 9 μέτρα, ενώ τα πιο σύγχρονα είναι από fiberglass. Η μεγαλύτερη περιφερειακή συγκέντρωση δείχνει ότι σε, σε αυτούς τους τόπους τα σκάφη είναι κυρίως ξύλινα 6 και 9 μέτρα και αυτά τα πέντε, αυτές οι πέντε περιφέρειες μαζί αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% του στόλου της αλίας μικρής κλίμακας. Σε αυτό το πίνακα, δεν ξέρω αν μπορείτε να τον διαβάσετε εύκολα από απόσταση, βλέπετε με κόκκινο είναι τα, πέντε πιο σημαντικά ε, πιο σημαντικές συγκεντρώσεις με ξύλινα και ε, ε, ε, fiberglass περιβλήματα των σκαφών που χρησιμοποιούν σειρώμενα δίκτυα. Εν συνεχεία έχουμε τις δράγες. Πάλι βλέπετε την κατανομή μεταξύ ξύλινων και πλαστικών σκαφών. Βλέπουμε επίσης τα σκάφη, τα αγριγρή, τα οποία είναι παλαιού τύπου αλίας, ξύλινα σκάφη και ούτω καθεξής η μεγαλύτερη συγκέντρωση είναι στα σειρώμενα και σταθερά δίκτυα. Πάνω από το μισό του ελευτικού στόλου χρησιμοποιεί αυτά τα, αυτόν τον εξοπλισμό και τα πάνω από τα μισά σκάφη είναι ξύλινα, ενώ τα σκάφη από fiberglass, με περίβλημα fiberglass, αντιπροσωπεύουν περίπου το 1 τρίτον. Ο πρόεδρος μας ζήτησε να ολοκληρώσουμε σε 20 λεπτά και Γι' αυτό σας συντομεύσω. Ποιε είναι λοιπόν, πού βρίσκονται οι μεγάλες πυκνότητες των σκαφών αυτών. Όπως βλέπετε από το χάρτη, είναι κυρίως στην Ελλάδα, Νότια Ιταλία, Νότια Ισπανία, Βόρεια Πορτογαλία και λιγότερο στην Εστονία και Νότια Φιλανδία. Το, δεύτερη πιο μεγάλη συγκέντρωση σκαφών 6 με 9 μέτρα ε, με παραγάδια είναι ε, Σαρδινία, Νότια Ιταλία, πάλι και Ελλάδα. Η πρώτη κατηγορία ήταν τα σειρώμενα σταθερά δίκτυα. Βλέπετε λοιπόν ότι η αλία μικρής ε, κλίμακας διανέμεται ας πούμε σχετικά ισόρροπα στην Νότια Ευρώπη, στις μεσογειακές παράκτιες χώρες και σε συγκεκριμένες περιοχές εντοπισμού. Δίνω πάλι το λόγο στον Γκρέαμ, ο οποίος θα μας μιλήσει περισσότερο για τον οικονομικό ρόλο της αλίας μικράς κλίμακας. Ευχαριστώ. Θέλω να τονίσω ότι υπάρχουν αντίγραφα της έκθεσης και περιλαμβάνουν πολύ περισσότερες πληροφορίες για τις ε, συγκεκριμένες τοπικές συγκεντρώσεις των σκαφών. Τώρα, μας ανατέθηκε επίσης η ανάλυση των οικονομικών και κοινωνικο-οικονομικών στοιχείων της αλλίας μικρής κλίμακας. Η συνολική αξία των αλλιευμάτων των εκφορτώσεων είναι περίπου 8 δις ευρώ και 26% ε, αυτής της ποσότητας ε, ε, προσφέρεται, εκφορτώνεται από την αλία μικρής κλίμακας. Η αλία μικρής κλίμακας απασχολεί 90.000 απασχολούμενους συγκεκριμένα έναντι 78.000 στον, ε, με τα, τα, σκάφη που είναι πάνω από 12 μέτρα και επίσης η αλία μικρής κλίμακας παράγει το 1 τρίτον των εκφορτώσεων ε, ανά άτομο όσον αφορά την προστιθέμενη αξία. Το 1 τρίτον της προστιθέμενης αξίας της αλίας παράγεται από τη μικρή κλίμακα. Ο περιφερειακός ρόλος, 20% των ΔΕΔΕΜΕ περιφέρειες ΝΑΤΣ 2 έχουν 0,1 ε, ποσοστό εξάρτησης ε, και αναλύσαμε την αγορά απασχόλησης, τα εισοδήματα κλπ. και μπορέσαμε έτσι να καθορίσουμε το βαθμό εξάρτησης από την αλία. Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανά σχέση απασχόλησης και η, όπως είπα, εξάρτηση αυτού του τομέα όσον αφορά η επίπτωση όσον αφορά την αγορά εργασίας εμφανίζεται σε αυτά τη στοιχεία βλέπετε ότι από τις 131 περιφέρειες, περιοχές μάλλον, 20 περιοχές ε, έχουν μια εξάρτηση από την αλία πάνω από 0,1%. Και, και το εισόδημα των εργαζομένων έχει μια εξάρτηση 0,05%, πολύ χαμηλή δηλαδή. Ε, πρέπει πρέπει να σκεφτούμε αυτά τα στοιχεία όταν συζητάμε την αξία αυτού του τομέα όσον αφορά την οικονομική του αξία, συγκρινόμενος με άλλες ε, οικονομικές δραστηριότητες. Οι περισσότερες περιφέρειες στην Ελλάδα είχαν την υψηλότερη εξάρτηση από την Αλία, πάνω από 1%, 8 τέτοιες περιφέρειες και 4 στη Γαλλία. Στις Περισσότερες ε, περιοχές υψηλής συγκέντρωσης, ε, ε, μικρής κλίμακας αλίας, έχει παρουσιαστεί μια μείωση της δραστηριότητα 10 με 30% τα τελευταία 10 χρόνια, ενώ οι περιφερειακές οικονομίες των ίδιων περιφερειών έχουν αυξηθεί κατά 30 με 60% στον αφορά το εισόδημα. οπότε βλέπετε ότι ο ρόλος των, ε, της αλλίας μικράς κλίμακας έχει σημαντικά μειωθεί την τελευταία δεκαετία. Αυτές, ε, αυτοί οι δύο χάρτες τώρα που βλέπετε δείχνουν ε, αυτά που σας παρουσίασε όσον αφορά την απασχόληση και την συγκέντρωση των απασχολούμενων στην Αλία στις διάφορες περιοχές που εντοπίσαμε. Ε, οι περιοχές αυτές, ΝΑΤΣ 2, είναι ακριβώς αυτές όπου η Ελία παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο σχετικά βεβαίως με τις άλλες δραστηριότητε. Αριστερά βλέπετε ότι η Ισπανία, Ελλάδα και οι βασικές περιφέρειες της Ελλάδας, όπως είπε ο Πάβελ, εκπροσωπούν τους, την υψηλότερη πυκνότητα όσον αφορά τους απασχολούμενους στην Αλία, μαζί με ορισμένες βαλτικές χώρες, μαζί με, ναι, ε, και αυτό, σας είπα, αυτή η ανάλυση επικεντρώθηκε στην ε, εξάρτηση της αγοράς εργασίας από την αλία. Σε σχέση βεβαίως με, άλλες, με άλλους τομείς απασχόλησης. Αν δείτε τώρα την εξάρτηση του εισοδήματος από την αλία, αυτό που είναι εντυπωσιακό σε σχέση με τον προηγούμενο πίνακα είναι σχεδόν ε, τέλεια εξαφάνιση των μαύρων περιοχών, δηλαδή των περιοχών υψηλής πυκνότητας. Δηλαδή βλέπετε εδώ περιοχές όπου η εξάρτηση από το εισόδημα δεν είναι μεγάλη. Ε, η εξάρτηση της αλίας όσον αφορά το εισόδημα είναι πολύ μικρότερη από ό,τι εξάρτηση από άλλους παραγωγικούς τομείς. Εδώ βλέπετε ακριβώς τον πίνακα των εξαρτήσεων. Βλέπετε την εξάρτηση του εισοδήματος ε, και την εξάρτηση της απασχόλησης στις περιοχές ΝΑΤΣ 2. Και από τον πίνακα αυτόν βλέπετε ότι λιγότερο από 5.000 άτομα απασχολούνται στην αλία μικρής κλίμακος σε περιοχές του ΝΑΤΣ 2 που έχουν πάνω από 1% εξάρτηση στην απασχόληση από την αλία. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Αυτή είναι η τελευταία μου διαφάνεια. Όπως σας είπα στην αρχή, το έργο μας δεν ήταν μόνο να παρουσιάσουμε στοιχεία για μια μακροσκελή ανάλυση πολιτικής, αλλά να δώσουμε την ευκαιρία της συζήτησης ε, των στοιχείων αυτών που συλλέξαμε και αναλύσαμε. Καταρχάς λοιπόν όσον αφορά τις ενδεχόμενες αλλαγές τους ορισμούς της αλίας μικράς, μικρής κλίμακας ε, έχουν γίνει, έχουν ακουστεί ορισμένες ιδέες ότι ίσως χρειάζεται μια αλλαγή της ορολογίας, μια αλλαγή του ορισμού για το τι σημαίνει small scale fisheries, SSF αλία μικρής κλίμακος. Επίσης ε, αυτό έχει άμεση επίπτωση και στην νομοθεσία. Ε, υπάρχουν διάφορες απόψεις και είναι σχετικό το ότι είναι μικρό. Μικρή κλίμακα. Ε, επίσης τα κριτήρια με τα οποία εμείς ορίζουμε εάν ένα αλλιευτικό σκάφος δείτε μικρό ή όχι. Και το πώς ορίζουμε τον εξοπλισμό. Δεν είναι εύκολο να πούμε ας πούμε ότι σε αυτή την περιοχή πυκνότητα, σε αυτή την περιοχή συγκέντρωσης θα εξαλείψουμε όλα τα σκάφη τα οποία έχουν χι διαστάσεις ή εξοπλισμό και θα τα εντάξουμε σε μια άλλη κατηγορία λίας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό έτσι αυθαίρετα. Ε, το, δεύτερο είναι ότι τα στοιχεία αυτά θα μας βοηθήσουν να μελετηθούν οικονομικές ε, αδυναμίες ε, και, οικονομική ισχύ, του τομέα αυτού. Ε, είναι πολιτικό το θέμα. Εάν θα συνεχιστεί, αν θα υπάρξει η συνέχεια της ενίσχυσης, της ανάπτυξης ή της υποστήριξης της αλληλίας μικράς, μικρής κλίμακας. Το θέμα εδώ είναι πολιτικό και άπτεται των γενικών πολιτικών ε, στόχων. Ε, δεν ξέρω ποια θέλετε, ποια ωφέλη θέλετε εσείς να ενισχύσετε περισσότερο και να τονίσετε ποιες αποφάσεις που θα πρέπει να λάβετε στο μέλλον. Αυτό έτσι ολοκληρώνω την παρουσίασή μου και δίνω το λόγο πίσω στην πρόεδρο και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και σχόλια. Ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις εξηγήσει που μας δώσατε σχετικά με την μελέτη. Είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα τώρα. Όπως και είναι το πράγμα όμως θα δώσω το λόγο στους ευρωβουλευτές τώρα προκειμένου να σας υποβάλουν ό,τι ερωτήσεις θέλουν για να διευκρινιστεί ακόμα περισσότερο αυτό το θέμα. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Ντέιβις είχε ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ναι. Όντως, πολύ βοήθησε η παρουσίαση αυτή. Πρώτη μου ερώτηση, λοιπόν. Μόνο στα αγγλικά υπάρχουν ε, οι παρουσιάσεις. Δώσατε τις πρώτες πέντε χώρες, ανάλογα με το μέγεθος του στόλου, αναχώρα. Δεύτερον, Ορισμός χρησιμοποιείται στο βασικό κανονισμό και πρόκειται για 12 μέτρα. Εσείς αναφερθήκατε σε ένα μέσο όρο 5 με 7 μέτρα. Οπότε τα 12 μέτρα πώς ε, φαίνονται, σαν βιομηχανικό σκάφος σε σχέση με αυτό που είπατε ότι είναι σαν μέσος όρος. Έπειτα, έχετε ανάλυση μήπως ε, τα σκάφη 10 με 12 μέτρων πόσο πολλά είναι και ποια είναι τα επιχειρήματα για να υποστηρίξουμε την άποψη ότι αντί για 12 μέτρα το όριο πρέπει να είναι 10. Λοιπόν, για να απαντήσω στο πρώτο σας θέμα, ναι, η έκθεση έχει διάφορα παραρτήματα που συμπεριλαμβάνουν όλα τα στοιχεία αναλυτικά και όχι μόνο αναχώρα μέλος όπως σας τα έδωσα εδώ, αλλά και βάσει των περιφερειών ΝΑΤ2. Οπότε εκεί όποιος ενδιαφέρεται θα βρει το μέγεθος των σκαφών όχι μόνο ανά χώρα μέλος αλλά και ανά σε κάθε χώρα μέλος. Για τη δεύτερη ερώτησή σας τώρα όσον αφορά το μέγεθος των σκαφών, το μήκος. Τα 3 με 5 μέτρα δεν αποτελεί κανένα μεσόρο. Πρόκειται για τα χαρακτηριστικά, τα κύρια του στόχου. Αλλά η έκθεση αναλύει τα νούμερα και συμπεριλαμβάνει τα, τον αριθμό των σκαφών ανάλογα με την κατηγορία. 3 με 6, 6 με 9 μέτρα κλπ. Τα στοιχεία δηλαδή στην έκθεση σας δίνουν τον αριθμό των σκαφών ανάλογα με το πόσα μέτρα είναι αναμέτρο. Δεν ξέρω αν απαντάω έτσι στην ερώτησή σας. Πρόεδρος, μια στιγμή να πάρουν όλοι το λόγο, έτσι μην αρχίσει ο καθένας από μόνος του να παίρνει το λόγο. Α κάνουν οι ευρωβουλευτέ όλες τις ερωτήσεις τους και μετά να απαντήσετε. Και κύριε Ντέβι, αν θέλετε, πολύ σύντομα σα δίνω το λόγο γιατί περιμένουν πολύ ακόμα. Ε. Τι θέλετε να ρωτήσετε. Και δώστε μας μια ιδέα παρακαλώ για το ποσοστό στο σύνολο του σκάφου. Ποιο είναι το ποσοστό των σκαφών 10 με 12. Και τι αλλιεύματα αλλιεύουν σε σχέση με το μέσο όρο. Ο κύριος Ρωμέβα τώρα. Ευχαριστώ. μετά τα τελευταία που άκουσα. Συμφωνώ ότι η αλλαγή του ορισμού για το τι είναι μικρής κλίμακα σκάφη θα ήταν κάτι χρήσιμο. Και γιατί πρώτα απ' όλα έχουμε ήδη αργήσει. Στο στάδιο που είμαστε έχουμε προσπαθήσει τον ορισμό αυτό να τον πετύχουμε ε, τελευταία στιγμή έτσι καλλιώς, πόσο μάλλον τώρα. Πάντως κάτι που ίσως θα ήταν ενδιαφέρον να συζητήσουμε είναι κάποια κριτήρια που να συνδέονται με συγκεκριμένες διαστάσεις και τις επιπτώσεις που έχουν αυτές στο περιβάλλον, για παράδειγμα, ή τον οποίον ο τρόπος αλίευσης πώς επηρεάζει. Άλλα κριτήρια δηλαδή, τα οποία να μπορούν να είναι χρήσιμα για να καθορίσουμε τελικά ποιος προχωράει σε πιο βιώσιμη αλία και ποιος όχι. Εσείς σκέφτεστε τη δυνατότητα αυτή να θέσετε και άλλα κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν. Ο κύριος Κάλαγερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συντάκτες της έκθεσης. Το πρώτο που πρόσεξα είναι ο αριθμός των απασχολούμενων σε στόλους κάτω των 12 μέτρων και ιδίω σε αυτούς που έχουν ξύλινα σκάφη 6 με 9 μέτρα. Είναι τρομακτικός αυτός ο αριθμός και εδώ τίθεται ένα τεράστιο θέμα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Όποιο τύπου γρηγρή και αν είναι αυτά, η απασχόληση σε αυτόν τον τομέα είναι τεράστια και προκύπτουν θέματα ασφάλειας των σκαφών αυτών το άλλο που πρόσεξα είναι 2,1 δισεκατομμύρια εκφορτώσεις από μικρούς τολίσκους, από μικρά σκάφη. Πολλές φορές ε, λοιπόν βλέπουμε τεράστιες ποσότητες να εκφορτώνονται ε, και πρέπει να τους συγχαρούμε για αυτή την προσπάθεια. Τρίτον, τα επιχειρήματα που υποστηρίζουν την αλληλεία μικρής κλίμακας. Δεν ξέρω αν είναι αντικειμενικά αυτά τα επιχειρήματα ή αν είναι υποκειμενικά και συναισθηματικά. Όταν σκέφτομαι την αλληλεία μικρής κλίμακας, αμέσως μου έρχεται κατά νου το, το θέμα του περιβάλλοντος. Είναι δικαιολογημένη μικρή αλληλεία από απόψεως περιβάλλοντος. Δεύτερον, όσον αφορά τις απορρίψεις, το, το ποσοστό των απορρίψεων που σημειώνεται από αυτή από αυτούς τους μικρούς τόλους είναι αμεληταίο. Αυτά είναι τα συν, αυτά είναι τα θετικά σημεία. Και το άλλο είναι η, η απασχόληση. Δεν, δεν έχει σημασία αν είναι τρεις ή τέσσερις εργαζόμενοι πάνω στο σκάφος. Η αλή αυτή είναι βασικά οικογενειακής φύσεως και έτσι επιβιώνουν οι οικογένειές τους. Ε, αυτά ήθελα να πω για να υποστηρίξω, για να δικαιολογήσω την, την στήριξη της αλίας μικρής κλίμακας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Γκάλαχερ και ευχαριστώ και τους συντάκτες αυτής ε, της ε, μελέτης. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε πολύ ε, καλά τα στοιχεία της αλίας μικρής κλίμακας, όπως ελέξη είναι κυρίως οικογενειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν εδώ και αιώνες και σε παράκτιες περιοχές. Και αυτές οι παράκτιες περιοχές είναι και περιοχές που συνήθως έχουν μία αδύναμη ε, υποδομή, μία αδύναμη ε, διάρθρωση Οπότε υπάρχει μία διασύνδεση πιστεύω μεταξύ ε, αδύναμων διαθροτικών στοιχείων και μικρής αλίας. Συνήθως αυτές οι περιοχές είναι και τουριστικές περιοχές. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε μία διασύνδεση μεταξύ της αλίας μικρής κλίμακας, των αδυναμιών των περιοφεριών αυτών και του ε, τουρισμού ε, για να δούμε ακριβώς πώς μπορεί να ε, βελτιωθεί η οικογενειακή απασχόληση. Πολλές φορές αυτή η οικογένεια απασχολείται ε, επί 24 ώρα συνεχή για να μπορέσει να επιβιώσει, για να διατηρήσει αυτή την, θα έλεγα, βιοτεχνική αλία. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η αλληλεία ε, έχει μεγάλη αξία και συνδέεται και με μία ε, παράδοση βιοτεχνίας αιώνων στο, στην Ήπειρό μας. Πρέπει να υποστηρίξουμε αυτούς τους ε, ήρωες, αυτούς τους εργαζόμενους σε αυτό τον τομέα διότι μεταδίδουν τις γνώσεις από γενιά σε γενιά, από πατέρα προς γιο, από οικογένεια προς οικογένεια. Και θα πρέπει να τους βοηθήσουμε να διατηρήσουν μία αηφόρο δραστηριότητα, ιδίως όταν βλέπουμε τι γίνεται στην αλία μεγάλης κλίμακας. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε τα πάντα να τα εξηγήσουμε επιστημονικά ή να εδραιώσουμε ένα μαθηματικό μοντέλο. Πολλά από αυτά είναι και ιστορικά γεγονότα υπάρχει ένα ιστορικό υπόβαθρο. Πάντοτε στις παράκτιες περιοχές η μικρή ελία έπαιζε ένα σημαντικό ρόλο και συνδέεται άμεσα και με τον τουρισμό ε, της περιοχής αυτής. Ευχαριστώ λοιπόν τους συντάκτες της μελέτης αυτές. Μας έδωσαν πολλές, ε, πολλά επιχειρήματα. Κυρία Λουβίν, Φερέιρα και Χίγινς. Και εκεί κλείνει ο κατάλογος των ομιλητών, Για αλλιώ δεν έχουμε χρόνο. Η κυρία Λεβίνη έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ τους συντάκτες για την παρουσίαση, ήταν σαφέστατη και πολύ ενδιαφέρουσα. Θα αναφερθώ στην οικονομική απόδοση. Η οικονομική απόδοση. Έχετε συγκρίνει την οικονομική απόδοση της μικρής αλίας έναντι της μεγάλης. Επίσης, έχετε καταγράψει την οικονομική απόδοση της αλίας ε, ε, μικρής κλίμακας σε σχέση με τον αλιευτικό εξοπλισμό και τους τρόπους που, που, που, που αλλιεύουν, τη μέθοδο αλίας. Τώρα, όσον αφορά τις επιδοτήσεις, έχετε μελετήσει την οικονομική απόδοση ε, σε σχέση με την επιδότηση, όταν το συγκρίνουμε αυτό δηλαδή με την αξία των εκφορτώσεων. Κύριος Φερέιρα. Δύο-τρεις παρατηρητήσεις και ερωτήσεις, αν μου επιτρέπετε. Θα ήταν χρήσιμο να έχουμε περισσότερη ενημέρωση για αυτή τη μελέτη πέρα από την παρουσίαση που μας έχει γίνει κυρίως όσον αφορά τη μεθοδολογία που, η οποία χρησιμοποιείται. Θα πρέπει να μπορούμε εμείς να αναλύσουμε και τη μεθοδολογία η οποία χρησιμοποιείται. Τώρα, όσον αφορά τον ε, ορίζοντα ο οποίος διαγράφεται ε, χρονικός, ε, τι είναι, είναι τα 10 χρόνια, τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας τα δεδομένα, ε, είναι 10 ετών παλιά. Από τότε υπήρχε μια εξέλιξη και ορισμένες χώρες μέλη κατά τη δεκαετία του 90 έχουν κάνει μεγάλες αλλαγές, ουσιώδεις, ενδεχομένως και αρνητικές όσον αφορά την ηλία. Γι' αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη, να λάβουμε υπόψη τη δεκαετία του 90, διότι ε, έχουμε απλώς μία, έτσι, ένα ορίζοντα χρονικό των 10 χρόνων. Ε, τα πράγματα προχωράνε. Θα θέλουμε να ξέρουμε δηλαδή πώς θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε, να δούμε πώς έχει εξελιχθεί ο τομέας αυτός. Έχουμε τα θέματα της ε, ε, απόδοσης αυτού του τομέα, τα θέματα που έχουν να κάνουν με την απασχόληση και κυρίως την απασχόληση. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι τα κριτήρια που χρησιμοποιείτε. Ε, αυσιρά κάνατε αντιμετώπιση του θέματος της απασχόλησης. Έχετε δει τα θέματα δραστηριοτήτων οι οποίες δεν είναι άμεσα ε, θέσεις εργασίας στην αλληλεία αλλά ε, συνδέονται σχετίζονται με το πριν ή μετά της ελίας. Έχουμε να κάνουμε και κατασκευή πλοίων, ε, ε, στη συνέχεια ας πούμε το πέρασμα των αλλιευμάτων. Θα ήθελα να πω να ξέρω με ποιο τρόπο βλέπετε το θέμα της αποσχόλησης. Και επίσης να πω και το θέμα της απόδοσης. Λάβατε υπόψη τις δραστηριότητες αυτές όταν μιλήσατε για την απόδοση της αλίας. Στην παρουσίαση υπάρχουν και κάποια σημεία τα οποία θα ήθελα να βαθύνω. Λέτε Φερρυπίν, εδώ και 10 χρόνια έχουμε μια μείωση, κάμψη, παρένθεση. Ε, η ανάπτυξη που μιλάτε έχει να κάνει με την αύξηση σε τόνους αλλιευμάτων. Ε, και στις περιφερειακά οι οικονομίες έχουν αναπτυχθεί 30-40%. Δεν ξέρω. Έχετε δεδομένα αναπεριοχή εγκεκριμένα ή έχουμε που πιστεύω εγώ δηλαδή διαφορετικές ε, καταστάσεις από χώρα σε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή μιλάμε για, γενικά για κάποιες, ε, κάποια δεδομένα ε, δείκτες οι οποίες όμως συγκαλύπτουν την πραγματική κατάσταση. Και φυσικά εδώ πέρα τι είμαστε σε κάποιο επίπεδο, έχουμε κάποιες, κάποια δεδομένα και τα οποία σημαίνουν κάτι και είναι σημαντικά. είναι όμως ε, δύσκολο να δει κανείς τι ακριβώς γίνεται από πίσω. Να δει κανείς τις επιπτώσεις της αλληλείας στις ε, παράκτιες περιοχές. Εδώ δεν είμαστε σε αυτό το πράγμα. Έχουμε δεδομένα που μας περνάνε σε ένα άλλο επίπεδο και το οποίο ε, συγκαλύπτει την κατάσταση. Αυτά σαν γενικές παρατηρήσεις. Θα ήθελα λοιπόν περισσότερη ενημέρωση για το έργο το οποίο έχει γίνει όσον αφορά τη μεθοδολογία η οποία έχει εφαρμοστεί. Σίγουρα αυτή η μελέτη είναι, θα είναι χρήσιμη για τις εργασίες μας, χωρίς αμφιβολία. Ήδη μας δίνει σημαντικές πληροφορίες. Πλην όμως θεωρώ ότι η μελέτη αυτή θα ήταν καλό να μας δώσει ακόμα περισσότερα στοιχεία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Higgins. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ε, παρουσίαση. Αλλά για μένα υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις στην έκθεση, γιατί εκεί που μιλάτε για την οικονομική και οικονομικοκοινωνική σημασία, λέτε ότι 90.000 απασχολούνται στη μικρή κλίμακα σαλία, ενώ 70.000 σε σκάφη πάνω από 12 μέτρα. Και μετά που μιλάτε για τις επιπτώσεις στην πολιτική, λέει ότι οι οικονομικές αδυναμίες της μικρής κλίμακας αλίας δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποστηρίξει η πολιτική μας μη βιώσιμες επιχειρήσεις. Η έκθεση όμως λέει ότι 90.000 απασχολούνται σε αυτήν. Οπότε αν 90.000 απασχολούνται εκεί, φυσικά και είναι βιώσιμοι. Οπότε τελικά ποιο είναι ο ορισμός της βιώσιμης αλίας. Επίσης, στην τελευταία σελίδα μιλάει για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μικρής κλίμακας αλίας. Πάλι αυτό σε συνδυασμό με τη βιωσιμότητα θέλω να το πω είναι, όπως είπαμε, μικρά σκάφη. Αλλιεύουν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. 80% των αλλιέων αλλιεύουν 10% των αποθεμάτων στα ευρωπαϊκά ύδατα. Και εγώ που είμαι Ιρλανδός σας λέω ότι πρόκειται κυρίως για περιοχές μακριά από το κέντρο, όπου η μόνη οικονομική δραστηριότητα εκεί είναι αλλία. Οπότε αυτό που θέλω να πω από τη δικιά μου την πλευρά ως Ιρλανδός είναι ότι οποιαδήποτε νέα κοινή ελευτική πολιτική πρέπει να λάβει υπόψη της το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι οι άνθρωποι που στη ζωή τους πρόσβαση μόνο στην αλία έχουν και δεν είναι δυνατόν να τους το απαγορεύσει αυτό η νέα κοινή ελευτική πολιτική. Έχετε το λόγο τώρα εσείς για να απαντήσετε στις ερωτήσεις που σας υποβλήθηκαν. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις και για τα σχόλια. Θα προσπαθήσω να απαντήσω κάπως σύντομα. 5.600 σκάφη είπαμε, τέτοια. Το άλλο που με ρωτήσατε για τα πολιτιστικά και περιβαλλοντικά ωφέλη. Αυτό δεν είναι κάτι μέσα στο πεδίο έρευνα που κάναμε εμεί. Εμεί ασχοληθήκαμε μόνο με την απασχόληση και το εισόδημα. Οπότε παρόλο που παρουσιάζουμε στοιχεία για το σε τι βαθμό ε, χρησιμοποιούν ε, τι τρόπους αλίας επιθετικές ή όχι, τα υπόλοιπα δεν ε, περιλαμβάνονται μέσα στο πεδίο της δικιάς μας έρευνας. Πρόκειται για μελέτη καθαρά για τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Στην έκθεσή μας επίσης περιλαμβάνουμε πληροφορίες για την οικονομική απόδαση του στόλου μικρής κλίμακας σε αντίθεση με εκείνους πάνω από 12 μέτρα. Την απασχόληση, προσθέμενη αξία κτλ. Και ο μικρός στόλος δίνει μεγαλύτερη ε, προσθέμενη αξία στην απασχόληση από ότι οι μεγάλες, ε, οι μεγάλες στόλοι βάσει της έρευνας CRD. Επίσης, ε, μιλάμε στην έκθεσή μας και για την επίδοση των ε, διαφόρων ε, ειδών αλίας που χρησιμοποιούν τα σκάφη αυτά. Δεν είναι δικός μας ρόλος να κοιτάξουμε τις επιδοτήσεις σε σχέση με τις ποσότητες των εκφορτώσεων, αλλά από άλλες αξιολογήσεις που έχουν γίνει από την Επιτροπή για την Κοινή Ελευτική Πολιτική, φαίνεται ότι οι επιδοτήσεις αποτελεί ένα δίκτυ εμείς όμως δεν το εξετάσαμε αυτό και κυρίως όχι για το στόλο μικρής κλίμακας. Μια άλλη ερώτηση που υποβάλλατε έχει να κάνει με την μεθοδολογία. Εμείς λέμε ότι μάλλον περιλαμβάνουμε στην έκθεση ολόκληρη τη μεθοδολογία. Υπάρχει δηλαδή πλήρης διαφάνεια για το τι μεθοδολογία ακολουθήσαμε, πώ αναλύσαμε τα δεδομένα και πώ καταλήξαμε στα συμπεράσματά μα. Όλα αυτά υπάρχουν στην έκθεση. Ε, δεν θα μπορούσα στην παρουσίασή μου να καλύψω όλες αυτές τις λεπτομέρειες γιατί μερικές φορές το μοντέλο που χρησιμοποίησαμε για να αναλύσουμε τα κλάστερς ήταν αρκετά περίπλοκο. Άλλη, η άλλη ερώτηση έχω να σας πω ότι ε, μας αποσχόλησε η οικονομική σημασία του στόλου μικρής κλίμακας αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Είδαμε όμως λιγάκι και τις τάσεις όσον αφορά τον αριθμό των σκαφών. Υπάρχουν λοιπόν στοιχεία για τις τάσεις στην έκθεσή μας, αλλά κυρίως αυτό που προσπαθούσαμε να κάνουμε είναι να δώσουμε μια εικόνα της σημερινή κατάστασης όσον αφορά το στόλο μικρής κλίμακας. Έρχομαι τώρα στην απασχόληση. Στόχος μας ήταν να κοιτάξουμε τι απασχόληση γεννούν τα σκάφη αυτά μικρής κλίμακας. Οπότε αυτό εξετάσαμε και δεν το είδαμε διαφορετικά. Ε, δεν εξετάσαμε το εισόδημα. Όπως ξέρετε, φυσικά έχει μεγάλη σημασία για πολλά σκάφη μικρής κλίμακας ανά την Ευρώπη. Ρωτήσατε επίσης κάτι για το κατά πόσο τα δεδομένα δίνονται αναπεριφέρεια. Ναι, στην έκθεση υπάρχουν λεπτομερείς πίνακες με όλες τις περιφέρειες NAT2. Με όλα τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, με όλους τους δείκτες, οπότε από εκεί μπορείτε να δείτε πόσο σημαντικό Εκεί είναι η στόλη μικρής κλίμακας στην κάθε περιφέρεια. Και έτσι έχουμε στο τελευταίο σας σημείο που έχει να κάνει με το κατά πόσο υπάρχει ε, δικαιολογία για τη συγκεκριμένη πολιτική όσον αφορά τα σκάφη μικρής κλίμακας. Κυρίως το πρόβλημα με τις μελέτες που κάναμε εμείς είναι ότι εξετάσαμε τις ε, περιφέρειες ΝΑΤΣ 2. Αν βέβαια αναλύσετε ακόμα περισσότερο σε τοπικό επίπεδο, ξέρουμε πολύ καλά ότι όντω η εξάρτηση όσον αφορά το εισόδημα και την απασχόληση σε άλλες μικρότερες περιφέρειες ή περιοχές είναι κάτι πολύ σημαντικό. Στην περίπτωση της Ιρλανδίας για παράδειγμα, εκεί έχει πολύ μεγάλη σημασία όντως ο στόλος μικρής κλίμακας για πολλές περιοχές εκεί. Στη μελέτη μας όμως δεν μπορέσαμε να κοιτάξουμε ε, θέματα που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό ή άλλα τοπικά ζητήματα, πολύ τοπικά που έχουν να κάνουν με την αλία μικρή κλίμακα εκεί. Όντω, αυτή είναι μια δυναμία της μελέτης μας, αλλά έπρεπε να δουλέψουμε με τους όρου αναφοράς που μας έδωσαν και με τα δεδομένα που είχαμε στη διάθεσή μας. Τέλος, για το κατά πόσο αιτιολογείται ή όχι μια συγκεκριμένη πολιτική. Εμείς προσπαθήσαμε στη μελέτη μας ε, να δούμε ότι αν υπάρχουν κίνητρα κοινωνικά ωφέλη και μπορείτε να πείτε ότι ναι, είναι πολύ σημαντική η μικρή κλίμακα αλεία, πρέπει να στηριχθεί. Αν όμω δείτε τον γενικότερο πίνακα και δείτε ότι δίνει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία η ε, αλεία μεγάλη κλίμακα, τότε θα καταλήξετε στο διαφορετικό συμπέρασμα. Οπότε εξαρτάται. Το κάθε είδο τόλου δίνει τα δικά του συν στην Αλία. Αν πρέπει να υπάρχει ειδική πολιτική για την μικρή κλίμακα αλία αυτό είναι ένα θέμα που αποφασίζουν οι πολιτικοί, όχι εμείς. Δεν ξέρω τώρα αν έχετε κάτι άλλο να πείτε, αν κάτι ξέχασα να απαντήσω. Ναι. Εγώ θα ήθελα ένα ακόμα στοιχείο να αναφέρω. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η μελέτη αυτή βασίζεται σε πολύ καλά παγιωμένα στατιστικά στοιχεία. Ιδίω από το Αρχείο Καταχώρησης Ελληνικού Στόλου της Κοινότητας. Το 95 ή 100% των στοιχείων αυτών είναι σωστό, διότι έχουν καταχωρηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Επίσης τα οικονομικά στοιχεία συλλέγονται εδώ και αρκετά χρόνια και πιστεύω ότι η ποιοτική διάσταση των συλλεξέντων στοιχείων είναι πολύ ισχυρή. Είναι δεδομένη και εγγυημένη. Άρα λοιπόν τα στοιχεία μας αυτά από στατιστικής άποψης είναι υγιέστατα. Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν υπάρχει άλλος που θέλει να μιλήσει. Ε, ολοκληρώνουμε εδώ τις ε, ερωτήσεις και απαντήσεις για τη μελέτη αυτή που υπάρχει σε πέντε γλώσσες. Εκεί είναι στη διάθεσή σας. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά και ιταλικά. Υπάρχει πλήρης έκθεση σε αυτές τις γλώσσες. Ωραία. Οπότε περνάμε τώρα. Τι έγινε, τι συμβαίνει. Στα πορτογαλικά δεν υπάρχει η μελέτη αυτή. Αργότερα, λέω, προς το παρόν σε πέντε γλώσσες. Αυτές που σας είπα. Μετά θα υπάρξει μελέτη και στις υπόλοιπες γλώσσες. Προς το παρόν υπάρχει μόνο σε αυτές τις πέντε. Συνεχίζουμε και δίνω το λόγο σε τρεις εκπροσώπους από διάφορες οργανώσεις διαφορετικών κρατών μελών που έχουμε προσκαλέσει εδώ για να μας δώσουν την άποψή τους όσον αφορά ε, τη νέα κοινή ελευτική πολιτική και που αυτή πρέπει να επικεντρωθεί. Δέκα λεπτά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ο κύριος Ομπράιαν από την Ιρλανδία. Έχετε το λόγο κύριε Ομπράιαν. Um, Ευχαριστώ. Το όνομα μου είναι Τζον Ομπράν και προέρχομαι από ένα, μια, ένα μικρό νησί και αντιπροσωπεύω τη μικρή νησιώτικη αλληλεία στην ε, παράκτια περιοχή του Ντόνεγκαλ στην Ιρλανδία. Ε, πριν ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούσε η αλληλεία αυτή εποχιακά και αλλήλευαν τα εποχιακά αλληλεύματα, ψάρια, αυστρακοειδή, αστακούς, καραβίδες κλπ. Από το 1972-73 ε, αναγκάστηκαν ε, να εφαρμόσουν τις διατάξεις της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό έχουν καταστραφεί οι ψαράδες και η αλία τους ε, σε αυτή την περιοχή και πιστεύω ότι φταίνε οι κοινοτικέ διατάξεις και ο τρόπος που έχουν ερμηνευτεί από την κυβέρνηση της Ιρλανδίας. Ειδικά η αλία της ε, Σαρδέλας ε, υπήρξε στην πελαγική αλία και του Σολομού στην αλία αναψυχής στα ποτάμια και στις λίμνες. Ο, επίσης απαγορεύτηκαν τα σειρώμενα δίχτυα στις ε, δυτικές ακτές της Ιλλανδίας και τις βόρειες ακτές της ε, Σκοτίας με τη δικαιολογία ότι δεν είναι καλό για τα λιεύματα, δεν είναι καλό για τις αγορές. Και αυτή είναι η παρούσα κατάσταση. Όσον αφορά την πολιτική, δεν έχουμε τα αριθμητικά στοιχεία για να ε, επιφέρουμε μια, διαφορά, μια, μια αλλαγή σε αυτή την κατάσταση. Έχουμε μόνο 67 ψήφους, η επαρχία του Ντόνεγκα δηλαδή, στις κοινοβουλευτικές εκλογές. Η φωνή μας λοιπόν είναι πάρα πολύ αδύναμη και γι' αυτό οι τοπικές ενώσεις ε, το, της μικρής αλίας ε, έχουν ενώσει τη φωνή τους με, άλλες, με άλλους συνεταιρισμούς ε, και προσπαθούμε να, να βοηθήσουμε την επιβίωση ε, μιας απασχόλησης η οποία πετελεί υψηλή δεξιότητα και είναι μια παραδοσιακή μορφή απασχόλησης. Ε, προσπαθώ να μιλήσω και αργά, λέει ο μιλητής, για να διευκολύνω τη διερμηνία. εμείς στον, στην στον οργανισμό μας εκπροσωπούμε ε, τους μικρούς αλληλείς ε, αλλά και συμμετέχουν μέλη μη κυβερνητικών οργανισμών. Ο στόχος της Ένωσης μας ε, είναι η εξασφάλιση της αηφόρου αλληλείας στα πλαίσια της κοινή αλληλευτικής πολιτικής της Ένωσης και η προώθηση των βέλτιστων πρακτικών. Επίσης, η εξασφάλιση της δίκαιης πρόσβασης στα αλλιευτικά ύδατα προς όφελος όλων των απασχολουμένων. Είναι αλλιευτική πολιτική δίνει ε, προτιμησιακή πρόσβαση σε συγκεκριμένες ε, περιοχές ε, αλίας και διακριτική μεταχείριση. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό που θα πρέπει να υπερισχύσει είναι η εξασφάλιση μιας αηφόρου πολιτικής. Ε, όπως αναγνωρίστηκε το 2010 από ένα ψήφισμα το οποίο πέρασε ε, ε, στην Ένωση και που λέει ότι η πρόσβαση στα γευτικά ύδατα δεν θα πρέπει να εξαρτάται μόνο από οικονομικά στοιχεία, αλλά θα πρέπει στην πολιτική αυτή να σωματωθούν και κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Αυτή όμως η χρήση εφαρμογή των κριτηρίων θα μπορέσει να οδηγήσει στην, ε, στο, σε ένα όφελος της αλληλείας, το να ωφελήσει η αλληλεία πιο απομακρυσμένες περιφέρειες και θα πρέπει επίσης να φροντίσουμε να γίνεται η αλληλεία με λιγότερο εντατικούς τρόπους, έτσι ώστε να έχει όσο το δυνατό χαμηλότερη επίπτωση στα τοπικά οικοσυστήματα. Και ε, μια άλλη παράμετρος είναι δημιουργία θέσεων απασχόλησης ε, και διατήρησης του κοινοτικού ιστού. Ε, έτσι θα μπορέσει η, αλία μικρής, η νησιώτικη αλία μικρής κλίμακας να προσφέρει ε, στην παραγωγή τροφίμων ε, αυτά όλα τα εξέσαμε στο σεμινάριο που έγινε, στην μερίδα εργασίας που έγινε στις Βρυξέλλες το 2010 για την αλία μικρής κλίμακος. όπου ακούσαμε τις εισηγήσεις ε, εμπειρογνωμόνων. Εμείς πιστεύουμε ότι πολλά ποιοτικά κριτήρια τα έχει αγνοήσει η Κομισιόν και δεν έχει προσδώσει την αναγκαία προσοχή στην παράκτια ανησιώτικη αλία. Έχει μάλλον περιθωριοποιήσει αυτή τη δραστηριότητα, διότι οι προτάσεις της ε, Κομισιόν ωφελούν κυρίως τους μεγάλους ε, ε, ε, αλληλείς, τις μεγάλες εταιρείες και τη βιομηχανική αλία. Αυτές οι μεγάλες αλληλευτικές εταιρείες έχουν ε, τη δυνατότητα να ψαρεύουν σε μεγάλη κλίμακα. Όμως ε, η μικρή αλληλεία έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει την αηφόρο ανάπτυξη της αλληλείας και την ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων. Έχουμε λοιπόν ε, αυτή, αυτή τη στιγμή με, μεγάλες απώλειες και 67% μειωμένο εργατικό δυναμικό στην αλία της περιοχής μας. Γι' αυτό ζητούμε από, την, από τα θεσμικά όργανα, όργανα να αλλάξουν τη ροή των γεγονότων και να αρχίζουν να εφαρμόζουν προγράμματα υφόρου περιβαλλοντικής ανάπτυξης, αηφορίας στην αλληλεία, ε, εύκολη πρόσβαση στις κατάλληλες αλληλευτικές περιοχές που προστατεύουν το περιβάλλον, ε, συμμόρφωση στους κανόνες, στους κοινωνικούς κανόνες ενίσχυσης ε, της τοπικής, των τοπικών δραστηριοτήτων, την παροχή μιας σειράς μέσων που θα δίνει τη δυνατότητα αλλιευτικών ευκαιριών με βάση τα κριτήρια αηφορίας και γενικώ ενίσχυση ε, και εφαρμογή πολιετών προγραμμάτων ε, με τα κατάλληλα μέτρα για να ε, εξασφαλίσουν τη συμμετοχή μικρών αλλιέων. Επίσης ζητούμε την εξασφάλιση της αηφόρου ανάπτυξης της αλληλείας με τη συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων παραγόντων και την καθιέρωση σαφών κριτηρίων και συνθήκων για να αποφευχθούν οι διαμάχες και οι αντιπαραθέσεις μεταξύ ενδιαφερομένων του κλάδου. Αυτό είναι το έγγραφο, μπορείτε να έχετε αντίγραφα. Τώρα έχουμε λοιπόν όλη αυτή την χιονοστιβάδα οδηγιών που έχουν καταστρέψει την αλία. Ίσως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πει τώρα ε, σε όλες τις κυβερνήσεις ότι θα βγάλουμε μία οδηγία η οποία θα ζητάει να σωθεί το πιο πολύτιμο είδος του πλανήτη μας, το άτομο, ο άνθρωπος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που τηρήσετε και το χρόνο σας. Ο κύριος Βαρτολομιέ Κοτσινιέ και έχει τώρα το λόγο. Πολωνία. Για 10 λεπτά έχετε το λόγο κύριε Μπαρτόλ Μιέιτς Κοστσίνιακ. ¿El representante polaco está aquí presente o es que no está? Tak, tak, już A, pardon, Szanowna pardon, Komisjo, dziękuję za możliwość wysłuchania publicznego. E, nazywam się Bartłomiej Goś... Δουλεύω για μια, ένα οργανισμό για αλληλείς και θα ήθελα να κάνω, κάνω μια παρουσίαση για την παραδοσιακή ε, αλληλεία στη Βαλτική. Τώρα, για τον ορισμό. Προετοιμάζοντας αυτή τη μελέτη, στηρίχθηκα στον ορισμό του κανονισμού που ορίζει ποια είναι η παραδοσιακή ελεία, για πλοία μικρότερα των 12 μέτρων που δεν χρησιμοποιούν μηχανέ. Αλλά στη βιβλιογραφία βρήκα και άλλα πράγματα. Άλλες πολύ ενδιαφέρον, άλλους ενδιαφέροντες ορισμούς ότι έχουμε να κάνουμε για, με μια αλληλεία η οποία διαφέρει πολύ από τη βιομηχανική διότι συρίζεται σε πολύ μικρότερα κεφάλαια ε, με εισοδήματα πολύ ταπεινά δυνατότητες οικονομικές πολύ μειωμένες περιορισμένες και λιγότερες ε, δυνατότητες στην, ε, το χώρο της εμπορίας αλλιευμάτων. Εμείς σαν οργανισμός παραγωγών, αναγνωρισμένος από τον Ιανουάριο, διαπιστώσαμε οι ίδιοι ότι έχουμε να κάνουμε ένα σημαντικό πρόβλημα. Ε, όταν κανείς έχει περιορισμένα μέσα οικονομικά, ε, αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες. Όπως και να κάνεις με, ε, με τα φράση, κάνεις αυτό το θέμα, ε, θα ήθελα εγώ να αναφερθώ κυρίως πώς έχει η κατάσταση. Σας δείχνω ξάλλου και μια φωτογραφία που βλέπετε, ένα, βλέπετε πλοία. Είναι δική μας ιδιοκτησία. Αριστερά Φερρυπίν, που βλέπετε αυτό κοτ 155. Μπορεί να αλλιεύσει μέχρι τα 5 μίλια. Για μια εβδομάδα ε, το, ο τζίρος που κάνει είναι 170 ευρώ. Ένα, όχι μάλλον, συγγνώμη, είναι το κέρδος. Αλλά απ' την άλλη πρέπει να δούμε ότι αυτή η αλληλεία παίζει ένα πολύ σημαντικό ε, ρόλο για την Πολωνία είναι σημαντική για την τοπική κοινότητα, για την Ήπεθρο. Έχουμε και την τουριστική δραστηριότητα, την ψυχαγωγία γύρω από αυτά και μπορεί κανείς να πει ότι η παραδοσιακή αυτή αλία αποτελεί μέρος του πολιτιστικού, θα λέγαμε, περιβάλλοντος, εικονιακών δραστηριοτήτων ε, στην Πολωνία. Και αυτό γίνεται επί αιώνες. Επίσης εδώ βλέπετε δύο φωτογραφίες με πλοία που είναι δικά μας. Πλοία 12 μέτρων το πολύ. Αριστερά βλέπετε ένα που είναι 9 μέτρα και 80 και το δεξιό ήταν 11 μέτρα και 80 καταστά. Έχουν κάποιες διαφορές, διαφοροποιήσεις όσον αφορά θέματα ασφάλειας το, ένα ας πούμε, το δεξιά πάει μέχρι 3,5 μίλια ναυτικά, ενώ το άλλο μπορεί να πάει μέχρι 12. Εδώ βλέπετε κάποιες άλλες φωτογραφίες. Τι βλέπουμε τώρα, εδώ έχουμε να κάνουμε πολιτιστική κληρονομιά. Πριν από 50 χρόνια, ε, με κουπιά. Για καμιά δεκαριά, ε, για δεκαετίες δεν είχε αλλάξει τίποτα. Εδώ βλέπουμε φωτογραφίες του σήμερα. Πλοία που χρησιμοποιούνται ακόμα. Και αυτά συγκρίνονται με, τα, με τις παλιές φωτογραφίες που σας είχα δείξει. Ε, η πολιτιστική διάσταση είναι σημαντική. Η παράδοση των αλλιέων έχει να κάνει με την εθνική διάσταση. Η παραδοσιακή αλληλεία τίνει να εξαλειφθεί και όλη αυτή η κληρονομιά. Γι' αυτό λοιπόν, για αυτή την αλία είναι σημαντικό να περιοριστεί η βιομηχανική αλία στη Βαλτική θάλασσα. Θα πρέπει να περιοριστεί η πρόσβαση στην παράκτης περιοχές ε, μεγαλύτερων πλοίων. Για τον σόλο τώρα τον πολωνικό μιλάμε για 789 πλοία τα πολλά από αυτά είναι ε, για παράκτη αλληλεία, δηλαδή μικρότερα των 12 μέτρων. Μετά από υπολογισμού του Εθνικού Ινστιτούτου, βλέπουμε ότι κάθε, κάθε, πλοίο, ε, κάθε πλοίο εξασφαλίζει 6 θέσεις εργασίας. Ε, ενώ κάποια άλλα μεγαλύτερα 10. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν επιπτώσεις όσον αφορά την παραδοσιακή και παράκτη αλία. Εδώ έχουμε να κάνουμε τεχνική του πλοίου, το μέγεθός του. Στην Πολωνία βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετά πλοία τα οποία είναι ξεπερασμένα και κοστίζουν πιο πολύ στη διαχείρισή τους. Ε, κατά μέσο, τα πλοία είναι, έχουν μέσο όρο ηλικίας 25 ετών και όπως καταλαβαίνετε ε, χρησιμοποιούν περισσότερα καύσιμα. Έχουμε τις εργασίες ε, συντήρησης της αιτήσιας Φερρυπίνου. Γιατί αναφέρω αυτά τα θέματα. Έτσι θέλω να αναφερθώ στην ε, μεταρρύθμιση που χρειάζεται να γίνει το θέμα της χρηματοδότησης των επισκευών των πλοίων. Χρειάζεται να γίνει εξυγχρονισμός σε αυτό το στόλο. Ε, οι εργασίες μπορούν να, να γίνουν με πλοία παλιά είναι να τα ξανακάνει κανείς ε, πιο σύγχρονα. Υπάρχει δυνατότητα από κοινού κάποιοι να αγοράσουν ένα καινούριο, μια μηχανή, καινούρια πλέον για να Εμείς μπορούμε να συγχρηματοδοτήσουμε τέτοιες δραστηριότητες και να συμμετέχουμε με ένα 40% του κόστους. Μετά έχουμε και την, ε, ε τις όπου εκεί πέρα υπάρχουν άλλα ποσοστά συγχρονατοδότησης. Θα πρέπει να δείτε αυτή τη διάσταση. Μήπως μπορεί η συγχρονατοδότηση να φτάσει στο ύψος του 80% ούτως ώστε να γίνει πιο επικερδής αυτός ο τομέας. Τώρα κάτι άλλο που μπορεί να έχει επιπτώσει στην αποδόση και την αποτελεσματικότητα του στόλου. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την υψηποδομέ στους, στους λιμένες. Στην Πολωνία έχει γίνει ένας εξυγχρονισμός πολλών λιμένων. Υπάρχουν επίσης υποδομές σε μικρά χωριά. Αλλά αυτό που αντιμετωπίζουμε σε γενικές γραμμές ε, ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των, ε, αυτής της υποδομής η οποία είναι ξεπερασμένη και αυτό ε, συμβάλλει στο να μην υπάρχει σωστή αποδοτικότητα. Έχουν εκφραστεί διάφορα αιτήματα που φτάνουν στον, στο ύψος των 500 εκατομμυρίων σλότη. εμείς ζητάμε και προσπαθούμε να γίνουν προσπαθήσεις ούτως ώστε να εξυγχρονιστούν οι μικροί λιμένες, χώροι ε, υποδομής, ε, όσο δυνατόν περισσότεροι στις υπάρχουσες ε, υποδομές. Τώρα, ε, η οικονομική διάσταση. Ε, εδώ έχουμε να κάνουμε τον εμπλωτισμό, θα λέγαμε, της δραστηριότητας αυτή, να δει κανείς όλη την αλυσίδα στο επίπεδο της αλίας. Η ανάπτυξη ζώνων αλλιευτικών επίσης να δοθούν δυνατότητες να ποικίλει το εισόδημα των αλλιέων για να μπορούν να εξασφαλίσουν καλύτερες προοπτικές. Ε, αλίευση, μεταποίηση και όλη η αλυσίδα μέχρι την τελική κατανάλωση του προϊόντος αυτό θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη βελτίωση της ε, αποδοτικότητας του τομέα αυτού. Έχουμε κάνει και αναλύσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Βλέπουμε ότι κατά μέσο ώρα ένα πλοίο έχει ένα καθαρό κέρδος 670 ευρώ εβδομαδίως με κάποιε βελτιώσει θα μπορούσαμε να φτάσουμε σίγουρα τα 800 ευρώ ανά εβδομάδα. Τώρα, πώ θα γίνει αυτό. Θα... Πέρασατε τα 10 λεπτά, ε. οπότε παρακαλώ ολοκληρώστε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Λοιπόν, κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στην ανάλυση που έχουμε κάνει δηλαδή ε, διασφάλιση της πρόσβασης και θέλουμε να δοθούν κίνητρα στους αλληλείς να οργανωθούν Θα πρέπει δηλαδή εδώ να δούμε το κανονισμό που αφορά την αλληλεία και εδώ να γίνουν κάποιες αλλαγές. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε ε, την πρόσβαση των αλλιέων σε τέτοιους οργανισμούς και επίσης να πω ότι θα δώσουμε μια έμφαση, πρέπει να δώσουμε μάλλον έμφαση. Ε, συγγνώμη, συγγνώμη, να προσθέσω λίγο ακόμα, κάτι ακόμα λέει ο μιλητής. Δηλαδή το θέμα που έχει να κάνει με την κοινωνική διάσταση. Αυτό είναι ένα σημαντικός παράγοντας για τους αλίες, τους παραδοσιακούς αλίες. Υπάρχουν κίνδυνοι για την ζωή τους, για την υγεία τους. Ε, διότι αντιμετωπίζουν και προβλήματα, είναι δύσκολο για αυτούς να περάσουν σε κάποια άλλη ε, επαγγελματική δραστηριότητα. Να τους δοθούν κινήτρα να μπορέσουν να επενδύσουν επίσης στην ε, τυποποίηση και μεταπόληση των αλλιευμάτων τους. Γενναίες και νεγές έχουν δραστηριοποιηθεί σε αυτό το τομέα η πρόσβαση σε οργανισμούς αλληλεγγύων λοιπόν θα ήταν κάτι πολύ θετικό. Ε, ε, σήμερα όπως έχει η κατάσταση οι αλληλείς δεν ενδιαφέρονται να ομαδοποιηθούν. Φυσικά ένας λόγος είναι ότι δεν υπάρχουν κεφάλαια. Όταν το θέμα της χρηματοδότης μπορεί να περάσει από 15 μέχρι 40% για τους νέους αλληλεί, ε, όταν ενδιαφέρονται να αγοράσουν ένα πλοίο εδώ υπάρχει διάσταση του, της οικογενειακής λέγαμε επιχείρησης. Επίσης η, τα προσόντα τους θα πρέπει να βελτιωθούν και μια ε, διαφοροποίηση στις δραστηριότητες. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη που πέρασα το χρόνο που μου είχατε στη διάθεσή μου. Σας ζητάω να τηρείτε το χρόνο σας για να σε βάρος των συναδέλφων σας. Τώρα έχει το λόγο ο κύριος Πλεσί ο οποίο εκπροσωπεί την γαλλική οργάνωση. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά παρακαλώ κύριε Πλεσί. Καλημέρα κυρία Πρόεδρε, κύριε και κύριοι. Εδώ θέλω να καταθέσω την εμπειρία μου από το 76 στη Βρετάνη. Έχω κάνει δύο παιχνιακές δραστηριότητες εγώ με, με τα χτένια από τον Οκτώβριο στον Απρίλη και επίσης με παραγάδια βυθού, ε, λαβράκι από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο. Αυτές οι δύο δραστηριότητες μου είναι ε, εποχιακές και χρησιμοποιούσα μόνο δύο μηχανές. Δράγα και παραγάδια βυθού. Και είμαι από τους τελευταίους που έχουν κάνει χρήση επιδοτήσεων ε, της Ευρώπης. Θα ήθελα να σας πω ότι η, η, μεταμορφ, η η αλλαγή που πρέπει να γίνει στην, ε, εδώ στι Βρυξέλλε, στην ε, Κομισιόν, είναι μια καταπληκτική ευκαιρία για να αντιμετωπίσουμε τα, τη νέα κατάσταση. Και ποια είναι τα σημαντικά σημεία για τη νέα πολιτική. Ε, παραδοσιακή αλία. Ποιο είναι ο ορισμό και ποια είναι η θέση τη στην κοινή αλληλευτική πολιτική. Η Επιτροπή είναι ξεκάθαρη. Ορίζει το μήκο των 12 μέτρων για να το ξεχωρίσει από τη βιομηχανική αλληλεία που φτάνει σε 100, γιγαντία πλοία των 135 μέτρων. Απ' την άλλη, έχουμε και τη μικρή δραστηριότητα αλληλευτική που με πλοία μέχρι 6 μέτρα. Η Επιτροπή στα κριτήριά της για τη λεγόμενη βιομηχανική ε, αλληλεία ε, συμπεριλαμβάνει όλα τα οποία έχουν να κάνουν με ε, κάποια δραστηριότητα χωρίς να λαμβάνει υπόψη το μήκος για παράδειγμα υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι, κάνουν, ε, ψαρεύουν απλάδια αλλά δεν αισθάνονται καθόλου ότι ασκούν μια ε, βιομηχανική αλία. Εμείς θεωρούμε ότι θα μπορούσε να μειωθεί το μήκος στα 13 μέτρα και επίσης να καθοριστεί και το, η δύναμη της μηχανής. Ποιες είναι οι, οι πτυχές τώρα. Όλα τα πλοία μικρότερα των 12 μέτρων, τα οποία ε, δραστηριοποιούνται σε ζώνες 12 ναυτικών μιλίων, ε, θα μπορούσαν να θεωρηθούν σαν τέτοια, όπου όμως ο ιδιοκτήτης είναι και αυτός στο πλοίο. Επίσης, ε, τα πλοία τα οποία αλλιεύουν και επιστρέφουν την ίδια μέρα στο λιμένι τους και πουλάνε το εμπόρευμα τους την άλλη μέρα. Και όλα τα πλοία φυσικά τα οποία σέβονται τη βιολογία των, των ε, ψαριών και τα οποία δεν αλλιεύουν σε περίοδο αναπαραγωγής. Απ' την άλλη, η μικρή δραστηριότητα, η ε, όπου ψαρεύει κανείς είδη τα οποία ε, βρίσκονται στην περιοχή ε, δεν έχει επιπτώσεις στην ανανέωση των αποθεμάτων. Αντιθέτως αντιμετωπίζει τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται με την υπεραλίευση, τη βιομηχανική. Για παράδειγμα βλέπουμε αυτοί που ψαρεύουν με καλάμι, με δράγα, έχουν χάσει 50% των δυνατοτήτων τους λόγω του ότι υπάρχει επιπτώση από τη μεγάλη και ανεξέλεκτη βιομηχανική ελία. Ε, μάθαμε φέρει πίν ότι ε, κάποιος θεωρούσε ε, μεγάλη δραστηριότητα ότι χρειαζόταν τέσσερις τόνους για να μπορέσει ε, να ψαρεύει, για να μπορέσει να πληρώσει μόνο τις φορές του προσωπικού του, του πληρώματός του. Να φανταστείτε ότι εγώ έχω ψαρέψει 4,5 τόνους σε 6 μήνες. Τώρα, ένα δεύτερο σημείο. Η απαγόρευση των απορρίψεων. Εδώ και δεκαετίες υπάρχει συνήθεια από τους ελείς να πετάνε ε, στους γλάρους ότι, ε, διάφορα είδη σε μεγέθους και ε, ψαριών τα οποία δεν είναι εμπορεύσιμα. Επίσης υπάρχει το πρόβλημα με τα δίχτυα και έχουμε ψάρια τα οποία δεν είναι ε, καταναλώσιμα. Αυτό σημαίνει ότι χαραμίζονται. Αλλά το θέμα είναι πώς κάνει κανείς σεβαστή την απαγόρευση. Δεν γίνεται να έχει κανείς μία κάμερα σε κάθε πλοίο. Θα πρέπει δηλαδή να κοιτάξουμε ούτως ώστε να γίνονται σεβαστοί κάποιοι κανονισμοί και να προστατεύονται οι γόνοι. Βλέποντας επίσης τη μείωση του προσωπικού, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μείωση και ελέγχων. Ε, εξάλλου με τα σημερινά πλοία μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούν να κρατήσουν όλα τα προσαπόρριψη ψάρια. Τώρα, ε, για τις ποσοστώσεις. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η βιομηχανική αλληλεία θα μπορούσε να διαχειριστεί το θέμα των ποσοστώσεων με κατάλληλο εξοπλισμό, διότι έτσι θα μπορούν να έχουν το κατάλληλο εμπόρευμα, το οποίο θα έχει μεγαλύτερη, μεγαλύτερη αξία στην αγορά και έτσι θα μπορεί να γίνει σεβαστή και η περίοδος αναπαραγωγή. Η Επιτροπή Περιφερειακή της Βρετάνης ζήτησε να γίνουν κάποιες αλλαγές και να γίνεται η καταμέτρηση όσον αφορά την ποσόστηση μετά την περίοδο ε, αναπαραγωγής. Τέλος η εμβάθυνση των ε, επιστημονικών στοιχείων. Θα πρέπει να γίνει μια πρόθεση προγράμματων τα οποία επιτρέπουν να έχουμε σωστά δεδομένα διότι τα λευτικά αποθέματα όπως ξέρετε δεν περιορίζονται σε μία θάλασσα. Εγώ θα ήθελα να σας πω εδώ πέρα επίσης και για μια μεγάλη αρχή θα πρέπει να είναι σεβαστή η βιολογία των ψαριών και κυρίως στην περίοδο αναπαραγωγής. Επίσης να έχουμε καθαρά νερά, χωρί λιπαγόνα ανθρώπινη προέλευσης, ένα καλύτερο θαλάσσιο οικοσύστημα, το οποίο βασίζεται στην ανανέωση των ε, αλληλευτικών αποθεμάτων. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μέχρι τις 5 και 10 τώρα θα έχουμε συζήτηση. Ο κύριος ε, Κάργη πρώτα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Από όλα αυτά που ακούσαμε, διαπιστώνουμε ότι η μικρή αλία, όπως συνηθίζουμε να τη λέμε, είναι πολύ σημαντική και είναι και αναγκαία. Πρέπει να τη στηρίξουμε. Πρέπει να τη στηρίξουμε διότι δεν είναι μόνο μια οικονομική δραστηριότητα, είναι συγχρόνως και κάτι που βοηθάει τη χωροταξία. Εμείς που ζούμε στις ακτές το ξέρουμε, χωρίς την μικρή Ελία δεν θα είχαμε λιμάνια. Από την άλλη όμως, νομίζω ότι πρέπει να αποφύγουμε μια παγίδα και αυτή είναι να βάλουμε από τη μια μεριά την μικρή αλία και από την άλλη μεριά τη βιομηχανική αλία. Τα δύο μοντέλα αλίας, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να συνεπάρχουν. Με ρύθμιση βέβαια και να ρυθμίσουμε ακόμα περισσότερο τη βιομηχανική αλία, το ξέρουμε, αλλά δεν πρέπει να τα βάλουμε αυτά τα δύο σε αντιπαράθεση, γιατί μπορούν να συνεπάρχουν και οι δύο μορφές αυτές αλίας, εφόσον οργανωθούμε καλά. Για άλλη μια φορά λοιπόν λέω ότι η μικρή κλίμακα αλεία και η βιομηχανική αλεία πρέπει και οι δύο να συνεχίσουν να ζουν. Βέβαια, στην νέα μορφή της κοινή ελευτικής πολιτικής, εισαγωγή ποσοστώσεων που μπορούν να μεταφέρονται, ίσως τελικά να θέσει σε κίνδυνο την μικρή αλία. Συμφωνούμε όλοι γι' αυτό. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι θέλουμε να διατηρήσουμε τον αριθμό σκαφών που έχουμε σήμερα στις ακτές μας. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Είναι επίσης αναγκαίο να καταγγείλουμε ό,τι και να συμβεί, οποιαδήποτε κατάχρηση λαμβάνει χώρο και να τις καταργήσουμε είτε πρόκειται για τη μικρή σκλήμα κασελίας είτε για την βιομηχανική. Γιατί και στη μικρή αλία δυστυχώς υπάρχουν ακόμα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν σέβονται τους κανόνες. Σε αυτούς πρέπει να επιβάλλουμε κυρώσεις. Όμως δεν νομίζω ότι πρέπει να δαιμονοποιούμε τον έναν ή τον άλλον. Γιατί πρέπει να στηρίξουμε και τα δύο είδη. Να στηρίξουμε την μικρή αλία, παρόλο που δεν την έχουμε καθορίσει επαρκώς. Λίγο πολύ ξέρουμε ποια είναι αυτή, αλλά όχι συγκεκριμένα. Εγώ πάντως εκεί θα ήθελα να μιζάρουμε στο να την ορίσουμε καλά. Ευχαριστούμε. Η κυρία Πάτκ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, εγώ θέλω να αναφερθώ στην ε, μικρή κλίμακα σαλίας, παρόλο που δεν έχω πολλά να προσθέσω σε αυτά τα τόσο καλά που ακούσαμε μέχρι τώρα. Κοιτάξτε, η μικρή αλία για μας εδώ στην Επιτροπή Αλίας είναι κάτι με το οποίο όλοι συμφωνούμε. Γιατί πολλές φορές μέχρι τώρα έχουμε πει πόσο μεγάλη σημασία δίνουμε σε αυτού του είδους τη δραστηριότητα. Το ακούσαμε και από τις μελέτες που παρουσιάστηκαν εδώ, ότι η μικρής κλίμακας αλία έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι είναι μια πρόσθετη αξία. Οι συνάδελφοι υπογράμμισαν και την μεθοδολογία, αλλά και την ακρίβεια των στοιχείων που έχουμε στη διάθεσή μας από την μελέτη που μας παρουσίασαν οι δύο κύριοι. Από όσα άκουσα λοιπόν, δεν συμπεριλαμβάνονται παρκώς οι άκρος απομακρυσμένες περιφέρειες, Αζόρες, η Μαδέρα, που είναι ευρωπαϊκή επικράτεια, αλλά που βρίσκονται πιο μακριά από το κέντρο, αλλά που έχουν ε, πολύ μεγάλη ακτογραμμή. Θα έπρεπε λοιπόν και αυτές να τις αναφέρουμε. Η μικρής κλίμακας αλία δεν χαίρει της ε, σημασίας και της προσοχής που θα έπρεπε να τις δώσουμε. Είναι πολύ πλοευρή η μικρή κλίμακα αλίας. Βασίζεται καταρχήν στον παραδοσιακό ε, τομέα. Ο τρόπος που γίνεται η αλία και ο τρόπος που φτάνει στο εμπόριο ε, το προϊόν της αλίας αυτής είναι ακόμα κάτι το παραδοσιακό. Και αυτό για μένα είναι μια προστιθέμενη αξία. Και γι' αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε όταν μιλάμε γενικά για την αλία. Με την μεταρρύθμιση αυτή που περιμένουμε και με τη μορφή που φαίνεται να έχει, αυτή η διάσταση δεν λαμβάνεται υπόψη όπως θα έπρεπε. για παράδειγμα, η σημασία που έχει η Αλία αυτή για την κοινωνική και την οικονομική διάσταση στις περιοχές όπου αυτή ασκείται. Όπως επίσης δεν λαμβάνουμε παρκώς υπόψη οικολογικά πόσο καλή είναι η μικρή αυτή αλία. Στην Επιτροπή Αλίας θα έχουμε σύντομα μια προφορική ερώτηση όπου εκεί θα αναφέρεται ακριβώς, ακριβώς αυτή η πολλαπλή διάσταση που έχει η μικρή κλίμακα σαλία. Θέλω να αναφερθώ και σε δύο ακόμα σημεία. Μιλάμε πάντα για την δραστηριότητα της αλίας που την κρίνουμε ανάλογα με την αυτονομία στη θάλασσα, τα σκάφη δηλαδή, με τον εξοπλισμό που διαθέτουν κλπ. Εγώ όμω πιστεύω ότι πρέπει να ξεφύγουμε τον παραδοσιακό αυτό ορισμό της αλίας μικρής κλίμακας. Σήμερα το πρωί ακούσαμε ότι δεν υπάρχει συμφωνία όσον αφορά για τον ορισμό της Μικρή κλίμακα αλεία και τη βιομηχανική αλίας, πώς δηλαδή ξεχωρίζονται οι δύο μεταξύ τους. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό, αλλά μια που συζητάμε αυτό το θέμα με τόσες λεπτομέρειες, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει κάποια συμφωνία όταν καθορίσουμε τα σκάφη που δραστηριοποιούνται στην μικρή αλία. Όπως είπαμε και πριν, είναι ένας τομέας με ιδιαίτερη αξία. Θα ξεκινήσουμε να αναλύουμε τα νομοθετικά έγγραφα της μεταρρύθμισης της κοινή ελευθερικής πολιτικής όπου να είναι και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι σε θέση να υπογραμμίσει τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε αυτού του τύπου αλλιές και αυτές τις δύο διαφορετικές ε, διαφορετικά ήδη σε Ευχαριστώ. Η κυρία Λουβένη. Ευχαριστώ πολύ όλους τους ομιλητές. Έχω ορισμένα σχόλια προς τον κύριο Μπράιαν, καταρχάς. Συμμερίζουμε την άποψη που εκφράσατε uh, Όσον αφορά τα ποιοτικά στοιχεία ε, των απόψεων σας. Σε αυτό συμφωνούν οι πράσινοι. Δεν είναι μόνο θέμα της ε, κατασκευής ή του μεγέθους, αλλά και του τρόπου αλίας. Αν είναι η μέθοδος αλίας αηφόρος ή όχι. Ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι ορισμένε μορφές αλίας μπορεί να βλάψουν το περιβάλλον. Δεν είναι λοιπόν εύκολο να βασίσουμε όλα τα κριτήριά μας σε κιλοβάτ, σε τονάζ ή σε ε, κατασκευή, σε διαστάσεις. Συμφωνώ επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, πρόσβαση κατά προτεραιότητα σε εκείνους που χρησιμοποιούν ε, σωστές περιβαλλοντικές και αηφόρες μεθόδους. Αυτό μπορούμε να το εφαρμόσουμε σε τοπικό επίπεδο και να δούμε πώς μπορούμε να διευκολύνουμε την πρόσβαση στις κοινέ ε, πηγές που είναι βεβαίως τα ψάρια, η αλία. Ε, όσον αφορά τώρα τα ε, άλευρα και τα άλλα παράγωγα προϊόντα της αλίας, εδώ υπάρχει μία διαμάχη που γίνεται βασικά στην περιοχή της Βαλτικής θάλασσας από πολιτικής άποψης πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα, όπως είπα, ε, σε αυτούς που αλλιεύουν και προσφέρουν ένα κοινωνικό όφελος. Να μην εξετάσουμε λοιπόν μόνο το ιστορικό υπόβαθρο των αλλιευμάτων και να δούμε αν έχουν γίνει παραχωρήσεις αλλίες ή όχι, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε την προαγωγή και ενίσχυση ε, αλλιευτικών δυνατοτήτων σε όσους κάνουν μια καλή δουλειά, χρησιμοποιούν καλές μεθόδους ε, και εφαρμόζουν κοινωνικά κριτήρια. Ο εκπρόσωπος ε, από την Πολωνία επίσης ανέφερε την διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων. Είναι σημαντικό σημαντικό αυτό για να μπορέσουμε να βρούμε ε, πρόσθετη, ε, προστιθέμενη αξία και να διαμορφώσουμε την αλή αυτή προσοδοφόρα, να μειώσουμε τους μεσάζοντες, να μελετήσουμε ε, την αγορά, τις αγορές, τυχόν ολιγοπολικές τάσεις ε, όπου οι αλληλείς αμείβονται ελάχιστα, μεσολαβούν οι μεσάζοντες και οι διανομής ε, έχουν μεγάλα κέρδη, ενώ ο ψαράς ε, επωφελείται ελάχιστα. Αυτά όλα πρέπει να καταπολεμήσουμε και αν επιτύχουμε θα ωφελήσουμε ιδιαίτερα την αλία στον τομέα της συγχρηματοδότησης και στην κατασκευή νέων σκαφών. Δεν το ευνοούμε αυτό. Δεν είμαστε υπέρ αυτού του μέτρου, διότι πιστεύω ότι έχουμε πλεονάζον δυναμικό στον ελιευτικό στόλο. Και πιστεύω ότι στο παρελθόν έχει εφαρμοστεί λάθος αυτή η πολιτική και δεν πρέπει να επαναλάβουμε τα λάθη. Ο κύριος Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω ε, τις εισηγήσεις που έγιναν και τους ομιλητές. Ευχαριστώ όλους όσους μίλησαν ε, και ως εκπρόσωποι της ε, αλίας μικρής κλίμακας και της παράκτιας αλίας. Εξ ονόματός τους ευχαριστώ και όλες τις οργανώσεις που εκπροσωπούν. Αναφερόμαστε εδώ σε έναν τομέα ο οποίος έχει συζητηθεί επιμακρών ε, στο Κοινοβούλιο. Μιλάμε για έναν τομέα ο οποίος τις τελευταίες δεκαετίες ε, είχε μία πάρα πολύ αρνητική εξέλιξη όπως ελέγχθη. Η κοινή αλευτική πολιτική, όπως είπε ο Ιρλανδός φίλος μας, ήταν καταστροφικός για την παράκτη αλία μικρής κλίμακας και τις παράκτιες περιφέρειες. Όχι μόνο στην Ιρλανδία, αλλά και σε άλλες χώρες. Είναι ε, ένα σημείο αυτό, είναι ένα γεγονός το οποίο δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε. Δεν αρκεί η ανάλυση της σημερινής κατάστασης μετά από αυτή την αρνητική συγκυρία δύο δεκαετιών ε, και να πούμε ότι δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα και τι μπορούμε να κάνουμε. Ε, δεν είναι σωστό αυτό δεδομένου ότι αυτή η κατάσταση διαμορφώθηκε υπό την ε, κάλυψη της κοινής αλληλευτικής πολιτικής η οποία αποδείχθηκε ότι ήταν καταστροφική για αυτού του είδους την αλία. Ε, πρέπει λοιπόν και να κάνουμε μία καταγραφή της σημερινής κατάστασης αλλά και να μελετήσουμε τη μελλοντική εξέλιξη. Ο φίλος μας από την Ιρλανδία μας ε, ε, παρουσίασε ένα μανιφέστο, μία δήλωση την οποία θέλει να την υπογράψουμε η οποία αναφέρεται κυρίως στους στόχους της αλληλείας αυτής και, των, και στις μελλοντικές εξελίξεις και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Ένα σημείο το οποίο συνεχώς τονίζουμε είναι να βελτιώσουμε την πρόσβαση στις πλουτοπαραγωγικές πηγές και να αξιολογήσουμε όλους τους τύπους της αλίας για να μπορέσουμε να προτείνουμε ε, αηφόρα μέτρα. Η αηφορία της αλίας είναι που μας ενδιαφέρει βάσει σωστών περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο για να επιβιώσει αυτή η αλία. Όμως η πρόταση της Κομισιόν δεν μας βοηθάει. Η Κομισιόν λέει στην πρόσβαση στις πηγές ε, βασίζεται ε, στα οικονομικά και χρηματοδοτικά κριτήρια. Ε, όλα βασίζονται στα οικονομικά κριτήρια. Όμως δεν είναι σωστό αυτό, διότι αυτό αντιτίθεται στους στόχους μας. Μάλιστα αντιτίθεται έντονα τα επιχειρήματα που παρουσιάστηκαν σήμερα δείχνουν ότι υπάρχει ένας εναλλακτικό τρόπος. Μία απομάκρυνση από αποκλειστικά οικονομικά κριτήρια και μία μεγαλύτερη, ένα μεγαλύτερο βάρος σε διαφορετικά κριτήρια. Η Πολλοί μας λένε ότι αυτό το ταμείο της αλίας ε, θα έχει ως στόχο την ενίσχυση και βοήθεια της μικρής αλίας. Δυστυχώς όμως δεν είναι αυτός ο τρόπος αυτό ε, που προτείνει η Κομισιόν, δεν είναι σωστές οι προτάσεις της Κομισιόν προς αυτό το τομέα. Θα ήθελα να σας δώσω μία συμβουλή. Βρισκόμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας και η Κομισιόν έχει παρουσιάσει τις νομοθετικές της προτάσεις που θα συζητηθούν στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο είναι μία διαδικασία η οποία θα κρατήσει αρκετούς μήνες. Και η συζήτηση που θα γίνει εδώ θα έχει μεγάλη σημασία για την εξέλιξη της διαδικασίας. Καθοριστική σημασία θα είναι η δραστηριοποίηση όλου το τομέα της, ε, μικρή, της αλλίας μικρής κλίμακος. Πρέπει να τους κινητοποιήσουμε, πρέπει να τους ενημερώσουμε και να δράσουν να αντιδράσουν στις προτάσεις αυτές. Πρέπει λοιπόν να οργανώσουμε ένα διάλογο και με τις εθνικές κυβερνήσεις και με τους τοπικούς παράγοντες και ενδιαφερόμενους ώστε να βρούμε ένα δρόμο διαφορετικό από αυτό που προτείνει η Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριος Γκάλαχερ. Ευχαριστώ. Ένα σχόλιο μόνο. έχουμε τρία άτομα εδώ οι οποίοι είναι πυρογνώμονες ε, στην Αλία και αντιπροσωπεύουν 90.000 εργαζόμενους. Αν το πολλαπλασιάσουμε αυτό επί τέσσερις, είναι περίπου 500.000 μισό εκατομμύριο άτομα, οι τρεις εκπρόσωποι της μικρής αλίας. Είναι σημαντικό λοιπόν να μην ξεχνάμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία αναγνώρισε τη σημασία της αλίας μικρής κλίμακας και παράκτιας αλίας. Και το ερώτημα στους ομιλητές είναι πιστεύουν ότι η αλία μικρής κλίμακας έχει επίπτωση στα αποθέματα και από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, οι απορρίψεις στα μικρά σκάφη είναι αρκετά χαμηλές. Αυτό σε τι οφείλεται, στο μικρό μέγεθος των σκαφών, στον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν, μήπως μπορούμε να συνάγουμε μαθήματα από αυτήν την πραγματικότητα. Ο κ. Γκρόβατσικ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, υποστηρίζοντας τις προτάσεις που έχουμε ακούσει και αυτά που μας είπε ο κύριος Φερέιρα για την κοινή αλλιευτική πολιτική ότι είναι ένα φιάσκο και ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί οριστικά, διότι δεν θα έχει κανένα θετική επίπτωση στην αλία. Σήμερα βλέπουμε το πρόβλημα της παραδοσιακής αλίας έτσι όπως διαγράφεται το θέμα και για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα αυτού. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα τομέα οικονομικής δραστηριότητας πολύ ευαίσθητο και όλοι νομίζω συμφωνούμε σε αυτό. Παρόλα αυτά, φαίνεται σημαντικό στα πλαίσια αυτής της κοινή αλληλευτικής πολιτικής να δούμε το θέμα της περιφερειοποίησης. Έχει εξάλλου ε, γίνει αναφορά σε αυτό. Ε, η Βαλτική Φερρυπίν είναι μια θάλασσα η οποία διαφέρει από τις άλλες θάλασσες. Η συνεργασία ανάμεσα στους τομείς, δηλαδή της βιομηχανικής αλληλείας και της παραδοσιακής, είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει κατανοητό. Υπάρχει μια αλληλεξάρτηση. Αυτό πρέπει να το δούμε και αλλού και σίγουρα η νομοθεσία αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί ε, σε άλλες ε, περιοχές θαλάσσιες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά επιμένω να το δούμε υπό την οπτική γωνία της περιφερειοποίησης. Είναι σημαντικό αυτό. Περιφέρειες. Δεν γίνεται αλλιώ. Η κοινή αλληλευτική πολιτική δεν μπορεί να πετύχει διαφορετικά. Τώρα, να δουν κάποια άλλη πτυχή του θέματος. Βλέποντας την ΚΑΠ, η οποία ε, δίνει διαφορετικές ε, ε, ε ανάλογα με τις ε, εδαφικές, τις ε, δυσκολίες, τις διαφορές αναπεριοχή, θα πρέπει να το δούμε και εδώ έτσι. Έχουμε το μεγάλο κόστος ε, το με το οποίο επιβαρύνονται οι φορολογούμενοι. Χρειαζόμαστε διατάξεις με διαφάνεια που δίνουν τη δυνατότητα να προστατευτεί η παραδοσιακή αλληλεία. Και τέλος το θέμα της νέας γενιάς η οποία δεν έχει καμιά δυνατότητα και καμία προοπτική θα λέγαμε για να δώσει μια συνέχεια σε μια φερρυπίν εικονιακή παραδοσιακή δραστηριότητα. Υπάρχει πολιτιστική δραστηριότητα της ε, αλίας. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιες δυνατότητες στα πλαίσια αυτής της κοινής αλληλευτικής πολιτικής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, έχοντας ακούσει τις παρουσιάσεις, θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχήν για αυτές. Συμφωνώ με αυτό που έλεγε νωρίτερα η κυρία Λέβεν για τις αγορές. Αν θέλουμε να ανταμείψουμε την βιωσιμότητα της παράκτιας αλίας και της μικρής αλίας, πρέπει να ψάξουμε να δούμε πώς ο καταναλωτής μπορεί να αναγνωρίσει τα αλλιεύματα που προέρχονται από αυτή την αλλία. με κάποιο είδους ετικέτες, σήμανση, δεν ξέρω. Το γράφω και στην εκθεσή μου. Πώς θα μπορέσει ο καταναλωτής να αντιληφθεί και να ανταμείψει την ε, αλία μικρής κλίμακας και τον μικρό όχι μόνο με τον ακούει ο μικρός Ελιάς ότι κάνει καλή δουλειά. Συμφωνώ με τόσα είπατε για την Ιρλανδία. Πράγματι και δεν ισχύει αυτό μόνο για την Ιρλανδία και δεν πρόκειται μόνο για τις οδηγίες για τους οικοτόπους. Τελικά είμαστε θύματα. Και μένα μου φτάνουν διαμαρτυρίες από μικρούς αλληλείς που μου λένε ότι έρχονται και τους λένε «Α, εμείς εδώ θα βάλουμε ανεμόμιλους ή εδώ θα βάλουμε ξέρω εγώ τι άλλο» ή ότι πρόκειται για μια μεγάλη περιοχή προστατευμένη χωρίς προηγουμένως να γίνεται καμία διαβούλευση. Οπότε τι κάνει ο κόσμος που ζει από την εκεί. Και πρόκειται, αυτό θέλω να πω, για μια προσέγγιση, για ένα σχεδιασμό από πάνω προς τα κάτω, χωρίς συνενώση, χωρίς διαβούλευση. Τους λένε αυτή την περιοχή σας την παίρνουμε. Εξαιτία σχεδίων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για παράδειγμα, ή για κάποιον άλλο λόγο. Πρέπει να αναγνωριστεί ότι πρέπει να γίνεται διαβούλευση με τον μικρό αλιά. Ότι η προσέγγιση πρέπει να είναι από κάτω προς τα πάνω και όχι ανάποδα. Και αν θέλουμε να ανταμείψουμε την μικρή κλίμακα αλία και τους μικρούς αλείς, να ξέρουμε ότι δεν πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση και ούτε η μεταρρύθμιση αυτή, έτσι όπως προβλέπετε, της κοινή ελευτικής πολιτικής θα βοηθήσει σε αυτό. Δεν πρόκειται να δείξει την αναγνώρισή μας στον μικρό αλία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακολούθησα με προσοχή όλη τη συνεδρίαση και ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Ε, θα είμαι εκείνη η οποία θα συντάξει το βασικό κανονισμό με τους συναδέλφους και έχω μία ερώτηση. Πιστεύω ότι θα ε, ε, ωφεληθούμε όλοι εάν στον κανονισμό βάσης περιληφθεί άλλο ένα κεφάλαιο ξεχωριστό με την αλία μικρής κλίμακας. Αυτή τη στιγμή αυτό δεν έχει συμβεί. Έχω πληροφορίες από την Κομισιόν ότι πολλά κράτη-μέλη πιστεύουν ότι δεν χρειάζεται αυτή η συμπερίληψη. Όμως εγώ πιστεύω μετά από το σημερινό απόγευμα ότι χρειάζεται απαραίτητο αυτό το κεφάλαιο και θα το προτείνω, το έχω συζητήσει με ορισμένους και ευχαριστώ και το ψήφισμα που έχω με στο τραπέζι μας σήμερα το απόγευμα. Πιστεύω ότι όλοι οι συνάδελφοι που συμφωνούν μαζί μου ε, να, να θέλουν ε, την προβολή της ε, και την προστασία της αλίας μικρής κλίμακας και πιστεύω ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να προστατεύσουν αυτό το τομέα όσο και να συζητάμε, όσο και να μελετάμε εδώ σε αυτό το σώμα, τίποτα δεν θα γίνει εάν δεν δεσμευθούν οι συνάδελφοι. Γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω τους ε, καλεσμένους μας. Σε μια συζήτηση έμαθα ότι οι ποσοστώσεις, εάν η διαχείρισή τους γίνεται εθνικά, σε εθνικό επίπεδο, μπορεί να ωφελήσουν για την βελτίωση των συντάξεων. Το έχετε συζητήσει αυτό ή είναι κάτι το αδιανόητο. Επίσης, ήθελα να σας ρωτήσω τι γνώμη έχετε για τα μακροπρόθεσμα προγράμματα διαχείρισης και άμα εξετάσω το, το MSY, πιστεύω ότι ε, έχετε πολλές γνώσεις που πρέπει να μας διαθέσετε, αλλά η μικρή αλία ε, δεν θα επαρκιέσει στο μέλλον. Χρειαζόμαστε και τη βοήθεια των επιστημόνων. Θα ήθελα να ξέρω πώς θα οργανώσετε αυτή τη συνεργασία. Δεν είναι σωστό εάν ε, κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Από τη μία πλευρά λέμε ότι θέλουμε να εφαρμόσουμε ε, τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια και από την άλλη ε, να κατηγορούμε το Natura 2000. Εάν δεν λάβουμε υπόψη τη βιοπικιλότητα, τα μέτρα προστασίας περιβάλλοντος, την ανάγκη προστασίας των ωκεανών, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά μέτρα διότι πριονίζουμε την καρέκλα πάνω στην οποία καθόμαστε. Ο κύριος Ντέιβις. Ευχαριστώ. Και εγώ υποστηρίζω την αλία μικρής κλίμακας. Ακούσαμε από τις ε, προηγούμενες εισηγήσεις την επίπτωση που έχει αυτός ο τομέας γενικά. Αλλά και οικονομικά οι επιπτώσεις είναι σοβαρές. Πολλοί ε, μικροί αλληλείς, αλληλείς δηλαδή μικρής ε, κλίμακας, δουλεύουν για ψίχουλα. Και είναι δύσκολο να, να, εξασφαλίσουμε την οικονομική τους επιβίωση. Είναι, είναι ελάχιστο το εισόδημα που έχουν Εάν, εφόσον λοιπόν ε, υποστηρίζουμε την αλία μικρής κλίμακος, αντί να κατηγορούμε συνέχεια την κοινή αλλιευτική πολιτική, ε, τις ποσοστώσεις, ε, τα επιτρεπόμενα αλλιεύματα. Ας κάνουμε επιτέλους κάτι για να προβάλλουμε την αλλία. Εγώ δεν βλέπω ε, μέτρα εφαρμόσιμα για την πρόθεση της αλλίας μικρής κλίμακος στην πρόταση της Κομισιόν, διότι η Κομισιόν με το πακέτο που μας παρουσιάζει λέει ειδικά ότι δεν ισχύει για την αλλία μικρής κλίμακος. Κάποιοι λοιπόν πρέπει να μου εξηγήσει γιατί. Οι αλληλείς όμως μικρής κλίμακος τι χρειάζονται για να επιβιώσουν και να βελτιώσουν την κατάστασή τους. Χρειάζονται ψάρια. Άρα λοιπόν πρέπει να μειώσουμε τις ποσοστώσεις ε, και τα αλλιεύματα των ε, βιομηχανικών στόλων. Και για να το επιτύχουμε αυτό θα έχουμε μεγάλες δυσκολίες, διότι οι μεγάλοι βιομηχανικοί στόλοι έχουν ισχυρές ομάδες πίεσης και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, ότι ο αγώνας είναι άνισος. Καλώς. Άλλο ένα νομίζω και μετά για να απαντήσετε οι τρει, Ο κύριος Ομπράιεν πρώτα να απαντήσετε. Δεν έχουμε άλλον βουλευτή τελικά, όχι. Παρακαλώ κύριο Ομπράιεν, ξεκινήστε εσείς να απαντάτε. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω για τον τρόπο που μπορούν να μειωθούν οι απορρίψεις και τι κάνουμε εμείς ε, στην Βόρεια Ιρλανδία αλλά και αλλού. Χρησιμοποιούμε διαφορετικά δίκτυα. Χρησιμοποιούμε διαφορετικά δίκτυα ανάλογα με το τι θέλουμε να πιάσουμε. Αν θέλουμε να πιάσουμε καλκάνι, χρησιμοποιούμε διαφορετικό μέγεθος ε, ματιού στο δίκτυ. Αν θέλουμε πέστροφα, κάτι διαφορετικό. Όταν μπορούσαμε ρέγγα να πιάσουμε, ε, πάλι χρησιμοποιούσαμε δίχτυα με μικρά μάτια που μόνο αυτό το ψάρι πιάναμε. Και ούτω καθεξής. Άρα, οι Ελλείς, από όπου και αν έρχονται, από τη Σκοτία, από την Ιρλανδία ή και αλλού, γνωρίζουν τι δίχτυ πρέπει να χρησιμοποιήσουν με τη μέγεθος ματιού. Έτσι διαχειριζόμαστε τα αποθέματά μας και έτσι αποφεύγουμε τις απορρίψεις. Και δεν είναι αδύνατον. Είναι πιο δύσκολο βέβαια με τις μηχανότρατες. Το καταλαβαίνω και στην Νότια Αγγλία, για παράδειγμα, που υπάρχει πολύ άμμος, ψαρεύουν και ήδη που δεν θα θέλαν. Είναι ένα δύσκολο πρόβλημα. Εγώ δεν έχω αλλιεύσει με αυτό το πρόβλημα, οπότε δεν έχω να σας προτείνω πώς να το κάνετε. Απλώς ξέρω, εμείς στην Ιρλανδία και η BMA, η οργανώση των αλλιών μας δηλαδή, τι κάνουμε. Φροντίζουμε, ακόμα και αν πιάσουμε ε, κατά λάθο ένα ψάρι που δεν θέλουμε, φροντίζουμε οι χρόνοι να είναι τέτοιοι που να μας επιτρέπουν να το πετάξουμε στη θάλασσα ζωντανό πάλι. Αυτό. Ε, Ευχαριστούμε, ο κύριος Βοτσινιάκ τώρα. Ευχαριστώ. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα στοιχείο μόνο. Εμείς είμαστε κατά του συστήματος που θα οδηγήσει στην εμπορία ακόμα πιο πολύ της αλίας. Δηλαδή ότι τελικά οι δυνατοί θα επικρατήσουν ενώ οι αδύναμοι θα εξαφανιστούν. Εμείς δεν θέλουμε αυτό το σύστημα. Προτιμάμε να κρατήσουμε το πάνω από 12 μέτρα χωρίς πρόβλημα. Καλά. Αυτό προτείνει η Επιτροπή. Δεν υπάρχει καινοτομία. Βλέπω ότι συμφωνείτε εσείς με την Επιτροπή τελικά. τέλο ο κύριος Πλεσή. Θέλω να πατήσω μόνο στον κύριο Ντέιβις. Παίρνω πάντα το... το χτένι. Σαν παράδειγμα. Εμείς ακόμα και για τα σκάφη κάτω από 12 μέτρα που είναι η ιδιαιτερότητά μας, χρησιμοποιούμε ένα μέσο το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα ότι τελικά οδηγούμαστε σε θάνατο της μικρής κλίμακας αλίας γιατί κατάσχεται όλο το προϊόν στο τέλος. Ευχαριστούμε. Δύο μου έχουν ζητήσει από το κοινό να πάρουν το λόγο. Αν είσαστε σύντομοι, πέντε λεπτά δηλαδή, ναι, ναι. Σα είδα, σα είδα. Μην σκόνετε τόσο πολύ το χέρι. Λοιπόν, δύο. Αν είσαστε σύντομοι και σε πέντε λεπτά τελειώσουμε για να περάσω στο δεύτερο πάνελ, έχει καλώς. Αλλιώς θα σας κόψω. Πρώτον, ο κύριος Τερίδης και μετά ο κύριος Λιμπεράτο. Ο πρώτος για τη Μεσόγειο και ο δεύτερος για τις Αζόρες. Δύο λεπτά ο καθένας το πολύ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουμε σε αυτήν ε, την ε, συζήτηση για τη νέα κοινή πολιτική. Θα σας πω πολύ γρήγορα ποιοι είμαστε και μετά θα σας δώσω και την άποψή μου για την πρόταση της Επιτροπής. Το Φεβρουάριο που μας πέρασε, εκπρόσωποι διαφόρων οργανώσεων ε, μικρής κλίμακας αλίας που έχω και μαζί μου εδώ από την Ελλάδα, από τη Γαλλία, τον Δημήτρη, τον Κρίστιαν, Συμβρεθήκαμε για να εντοπίσουμε προβλήματα και να ανταλλάξουμε απόψεις. Με διάφορες οργανώσεις λοιπόν, ε, από την Μεσόγειο πρώτα απ' όλα, και ένα από τα θέματα στο οποία συμφωνούμε είναι ότι πρέπει να διαρθρωθεί η διαχείριση και να γίνει κοινή. Δεν μπορεί ένας να επικρατεί. Χρειάζεται λοιπόν διαβούλευση για την κοινή ελευτική πολιτική. Παρ' όλα αυτά το στοιχείο αυτό το άφησε απ' έξω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι δεν έλαβε υπόψη στα συμφέροντα της μικρής κλίμακας Η διαχείριση μπορεί να γίνει με προγράμματα βιωσιμότητας του τομέα, διασφαλίζοντας την ακυρότητα των πόρων και την επιβίωση της δραστηριότητας αυτής μακροπρόθεσμα. Η συνδιαχείριση έχει σαν αποτέλεσμα ότι συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι και ενδιαφερόμενοι στα προγράμματα διαχείρισης και ενισχύεται αυτό από το γεγονός ότι και τα θα είναι πιο σταθερά και λαμβάνουμε υπόψη μας τους χώρους αλίευσης, όπως επίσης και τις προστατευμένες περιοχές. Ήδη από το 15ο αιώνα έχουμε ξεκινήσει να έχουμε συνδιαχείριση των ε, περιοχών αλίευσης. Εμείς ήδη οι αλίες το θέλουμε αυτό γιατί έχουμε εμπειρία το τι γίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο και ξέρουμε ότι έτσι έχει βελτιωθεί η κατάσταση των αποθεμάτων και η κατάσταση των ίδιων των ε, αλλιέων. Το λέει αυτό και ο επιστημονικός κόσμος, ότι η συμμετοχή βοηθάει και ότι έτσι θα επιβιώσει καλύτερα ο τομέας και θα γυριστούμε καλύτερα τους πόρους. Η μικρή κλίμακα σαλή ζητάμε να αναγνωριστούμε σαν μέρος της διαχείρισης του περιβάλλοντος και έτσι θα μπορέσουμε να δραστηριοποιηθούμε στην εκπόνηση πολιτικών για την διατήρηση των πόρων. Συγγνώμη, ξέρω ότι έχει λήξει ο χρόνος μου, αλλά να, τι θέλω να πω, ότι εμείς δεν συμφωνούμε με αυτά που λέτε για την ε, Μεσόγειο και για την πρόταση για τις απορρίψεις. Πιστεύουμε ότι δεν θα αποφεληθούμε. αλλά θα αλλιευθούν ήδη, τα οποία έχουν να κάνουν με τη βιομάζα πιο πολύ. Η δικιά μας πλαταφόρμα πάντως δεν θα σταματήσει τη δουλειά μας, δεν θα σταματήσουμε στην μεταρρύθμιση γιατί ό,τι και να γίνει θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε ώστε οι κοινότητες των αλλιών μας να εξακολουθούν να ζουν και να προστατεύουν μια κληρονομιά που και πολιτιστικά και περιβαλλοντικά είναι αξιοσημείωτη. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Λιμπεράτο τώρα και σας παρακαλώ δύο λεπτά ακριβώς για να περάσουμε στο δεύτερο πάνελ, παρακαλώ. Είμαι από την Πορτογαλία. Είμαι ο κύριος Λιμπεράτο, θα είμαι σύντομος. Ένα μόνο ερώτημα. Εδώ και 9 μήνες συζητήσαμε για την μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και έχουμε εμπιστοσύνη προτάσεις για τις αλλαγές. Περιμέναμε. Όλα τα είδαμε όμως το σύνολο του κανονισμού μας προτάθηκε, όλες οι προσδοκίες μας έσβησαν, χάθηκαν. Ελπίζουμε λοιπόν, λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων του, να κάνει το ίδιο προτάσεις, να κάνει κατάθεση τροπολογιών σε σχέση με τις προτάσεις της Επιτροπής και να μπορέσει ούτως ώστε ε, να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη μας, διότι το πρόβλημα που υπάρχει σήμερα στον χώρο των αλλιέων είναι το θέμα της εμπιστοσύνης. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη, ειλικρινά. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει μια μεταρρύθμιση της κοινής αλλιευτικής πολιτικής. Γι' αυτό εσείς είσαστε αυτοί που θα δείξετε στον τομέα της αλλιείας ε, ότι μπορούν όντως να γίνουν κάποιες αλλαγές. είχε γίνει συζήτηση στην Πράσινη Βίβλο. Τότε είχαμε ακόμα εμπιστοσύνη. σήμερα τη χάνουμε όμως. Ελπίζουμε όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαν τέτοιο που είναι και οι δυνατότητες που έχει να μπορέσει ε, στα πλαίσια της συνθήκης του, της Λισαβόνος να μπορέσει να κάνει κάτι και να ξανααποκτήσουμε, να ξαναέχουμε εμπιστοσύνη. Ε, segundo panel, que es más de lo mismo, estaría... Πρώτο πάνελ έχει τελειώσει. Τώρα θα περάσουμε στο δεύτερο, το οποίο έχει να κάνει με το ίδιο θέμα, αλλά θα δώσει έμφαση περισσότερο στο τι ακριβώς είναι αυτή η μεταρρύθμιση. Στο δεύτερο πάνελ θα δώσω το λόγο για 10 λεπτά στο... στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Ερνέστο Πένας θα θα μιλήσει εκ μέρους της Επιτροπής λοιπόν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, για να αρχίσω θα ήθελα να επανέλθω σε αυτά που είπα το πρωί, ότι η αλία μικρής κλίμακας, ε, όπως και σε άλλους τομείς, απασχολεί την Κομισιόν ιδιαίτερα επειδή έχουμε αναγνωρίσει ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα από την εποχή της αρχικής πρότασης και την πράσινη βίβλο. Έχουν λοιπόν αλλάξει τα πράγματα από τότε μέχρι τις σημερινές προτάσεις. στο νέο έγγραφο, στο, στο, στην πράσινη βίβλο η Κομισιόν έδειξε σαφέστατα πόσο σημαντική είναι η αλία και τότε προτείναμε ε, ότι η αλία μικρής κλίμακας όχι μόνο είναι σημαντική, αλλά και... Ε, Θέλαμε ένα ειδικό ε, καθεστώς. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η ανησυχία υπήρχε έτσι κι αλλιώ στην Πράσινη Βίβλο. Στη συνέχεια βέβαια είχαμε κάποια εξέλιξη και όπως συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις με τη μεταρρύθμιση, το ξέρουμε πολύ καλά, είναι ένα από τα θέματα για τα οποία πολλοί από εσά και τα κράτη-μέλη μας λένε ότι η πρόταση δεν αντιστοιχεί ακριβώς στο επίπεδο αποδοχής που αναφέρει η Πράσινη βίβλο. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό. Όταν εμεί μιλάμε για ένα μικρό καθεστώς για την μικρή αλία, μιλούσαμε για δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα για τη δυνατότητα ενός καθεστώτος διαχείρισης χωριστό με τα δικά του μέσα και μιλούσαμε βέβαια και για την δυνατότητα καθορισμού ενός καθεστώτος ειδικού ενισχύσεων στον τομέα. Αυτό στα πλαίσια της διαφορετικής μας πολιτικής. Το αποτέλεσμα μετά από τις ε, διάφορες διαβουλεύσεις που κάναμε καταλήξαμε στο εξής όσον ε, αφορά την ε, στήριξη. Η ειδική στήριξη στη μικρή αλία είναι κάτι με το οποίο όλοι συμφώνησαν. Κανείς δεν είχε αντίρρηση στο να υπογραμμίζεται ιδιαίτερα η μικρή αλία. Όμως, όσον αφορά τη δυνατότητα κάποιου χωριστού καθεστώτος δεν υπήρχε ξεκάθαρη ιδέα. Οπότε τελικά αυτό που προτείνει η Επιτροπή στον κανονισμό που έχετε για ένα νέο βασικό κανονισμό, έχετε κάποια, αλλά όχι πολλά στοιχεία διαφοροποίησης, πώς διαφοροποιείται δηλαδή η μικρή αλία από την άλλη. Και θα αναφερθώ εδώ σε κάποια στοιχεία που ίσως, εδώ έτσι καλώς σας μιλάω και κάτι προετοιμάζουμε ακόμα, ίσως βρείτε στον τελικό κανονισμό. Και θέλω να κάνω μια διαφοροποίηση εδώ που είναι σημαντική. Τι έχουμε στο βασικό κανονισμό. Όπως γνωρίζετε, έχουμε στην πράξη μία μόνο διάταξη η οποία διακρίνει την μικρή αλία από τις άλλες και είναι εκείνη που έχει να κάνει με την εφαρμογή συστημάτων επεξεργασίας στα σκάφη που είναι πάνω από 12 μέτρα. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο στοιχείο που διαφοροποιεί τη μικρή αλία από την άλλη. Ήδη εδώ η Κομισιόν πολύ γρήγορα μας το έδωσε αυτό στις διαβουλεύσεις. Μας το είπε από την αρχή ξανά και ξανά ότι το σύστημα αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα μια υπερβολική συγκέντρωση στα χέρια των μεγάλων σκαφών σε σχέση με των μικρών. Και είπαμε ας προτείνουμε αυτό τον μηχανισμό, αλλά ας βγάλουμε από εκεί την μικρή αλία. Και αυτό όχι γιατί πιστεύουμε ότι η ρύθμιση είναι κακή, αλλά γιατί από τη διαβούλευση καταλήξαμε στο ότι οι μικροί κινδυνεύουν. Κινδυνεύουν τα δικαιώματά τους στην αγορά και σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλύτερο να υπάρχει εξαίρεση. Αλλά υπάρχουν εδώ δύο ακόμα στοιχεία σημαντικά. Για παράδειγμα, το θέμα των 12 ε, μιλίων. Αυτό είναι κάτι ξεχωριστό από την ε, μικρή αλία. Όσοι θέλανε να το επεκτείνουν αυτό που ήθελε και η Κομισιόν, είναι γιατί καταλάβαμε ότι τα 12 μίλια έμεσα είναι ένα μέσο από το οποίο ευνοείται η μικρή αλία. Υπάρχουν εδώ όμως και άλλα στοιχεία πολύ σημαντικά. Στην συζήτηση αυτή φάνηκε ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον. Ακούστηκαν πολλές απόψεις. Κατηγορείται την πρότασή μας. Όμως ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί διαπιστώσαμε ότι πολλές από τις διαμαρτυρίες που μας έρχονται από τη μικρή αλία στην πραγματικότητα είναι διαμαρτυρίες που έχουν να κάνουν με τις εθνικές ρυθμίσεις, με την εθνική διαχείριση να το πω πιο σωστά. Το είπαμε και το πρωί και το ξαναλέω τώρα η κοινή αλληλευτική πολιτική βάζει ποσοστώσεις. Από εκεί και πέρα, ανάμεσα στα διάφορα είδη, στα διάφορα τμήματα της αλίας, είναι τα κράτη-μέλη που κάνουν ε, το χωρισμό. Άρα μέσω εθνικών πολιτικών θα μπορούσε να λυθεί αυτό το πρόβλημα και σήμερα και στο μέλλον. Μια διάσταση λοιπόν πολύ σημαντική που θέλω να υπενθυμίσω γιατί πολλές φορές τα βάζουμε με την κοινή ελευθερική πολιτική ε, για πράγματα τα οποία είναι εθνική αρμοδιότητα. Τώρα, κυρία Πρόεδρε, όσον αφορά το μελλοντικό δημοσιονομικό κανονισμό, εδώ επιτρέψτε μου να σας δώσω κάποιες ενδείξεις για το τι μπορεί να περιλαμβάνει ο κανονισμός αυτός. Η πρόταση, όπως σας είπα, βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας, οπότε δεν μπορώ να ξέρω πώς θα έχει στο τέλος, αλλά επειδή θέλω να υπάρχει διαφάνεια, προσπαθώ να σας πω όσο γίνεται περισσότερα από αυτά που ξέρω, από τις ενδείξεις που έχω για το πώς θα έχει η ρύθμιση αυτή. Βέβαια, ε, προσοχή, όσο δεν έχει εγκριθεί 30 Νοεμβρίου από τους Επιτρόπους, μην το θεωρήσετε σαν κάτι δεδομένο, σας το λέω με κάθε επιφύλαξη. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα στοιχεία τα οποία εμείς εξετάζουμε. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα βασικό θέμα και αυτό είναι ότι ανάμεσα στα διάφορα κριτήρια τα οποία θα προτείνει η Κομισιόν για την κατανομή των πόρων μεταξύ των κρατών μελών, ένα από τα κριτήρια μπορεί να είναι το βάρος του παραδοσιακού τομέα στο κάθε κράτος μέλος. ακριβώς για να μην ζημιωθεί η παραδοσιακή έλεια. Υπάρχει ένα δεύτερο στοιχείο σημαντικό και αυτό είναι το εξή. Στις αποφάσει δεν μπορώ να σας δώσω βέβαια νούμερα γιατί αυτά τα συζητάμε ακόμα, αλλά κατά πάσα πιθανότητα στην πρόταση θα γίνεται ειδική μνήμα στην ε, ένταση της βοήθειας για την μικρή αλία. Προσπαθούμε δηλαδή να φτιάξουμε ένα σύστημα που θα υπάρχει ένα ποσοστό κοινοτικής παρέμβασης και, τον ε, και του δημοσίου που θα εφαρμόζεται γενικά, αλλά για την μικρή αλία το ποσοστό θα είναι μεγαλύτερο. Για να το πω αλλιώ. Άλλη ιδέα που εξετάζουμε. Ο βαθμός της οικονομικής ενίσχυσης να είναι μεγαλύτερη για την μικρή αλία από ότι για άλλα προγράμματα που συμμετέχουν ε, και άλλα τμήματα του ελευτικού στόλου. Κάτι άλλο στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι το X4. Εδώ υπάρχει ένα θέμα μικρής αλίας, το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με την μικρή αλία. Είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με την διατήρηση των παράκτιων κοινοτήτων που εξαρτώνται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από τις αλληλευτικές δραστηριότητες. Άρα, όταν θέλουμε να προστατεύσουμε την μικρή αλία, δεν μιλάμε μόνο για τα σκάφη, μιλάμε για τους ανθρώπους. Σήμερα το πρωί το ξαναείπα, το είπε και η Επίτροπος, ότι στα πλαίσια αυτά θέλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη όθηση στην αντιστοιχεία αυτού που σήμερα είναι ο άξονας 4. Η οικονομική διαφοροποίηση, δηλαδή η πρόθεση των συμπληρωματικών στην αλληλεία δραστηριοτήτων. Και παρόλο που δεν λέγεται ότι πρόκειται για τα σκάφη κάτω των 12 μέτρων, ε, περί αυτού θα πρόκειται. Στόχος είναι να ενισχύσουμε οικονομικά τις περιοχές αυτές που εξαρτώνται περίπου αποκλειστικά από την αλία, δηλαδή την μικρή αλία. Θα δούμε αν τελικά έτσι εγκριθεί από την Κομισιόν. Αν ναι, νομίζω ότι αυτό θα έχει μεγάλη σημασία. Θέλω επίση να σας πω ότι ένα από τα στοιχεία που θα συμπεριλαμβάνονται στο δημοσιονομικό κανονισμό και που δεν θα αφορούν μόνο την μικρή αλία, είναι πράγματα όμω από τα οποία έχει να υποφεληθεί η μικρή αλία, μια από αυτή χρειάζεται τέτοιου είδου βοήθεια, είναι επειδή είναι ευάλωτη και οικονομικά και από πλευρά διαχείριση η αλία αυτή, να γίνεται μια διαφοροποίηση στην αγορά των προϊόντων που μας έρχονται από την μικρή αλία. Με το καθεστώ ενισχύσεων Βέβαια δεν θα περιοριστούμε στην μικρή αλία, αλλά η μικρή αλία έχει να κερδίσει περισσότερο. Αυτή είναι που μπορεί να υποφεληθεί περισσότερο από μια τέτοια διάταξη. Το ίδιο και για τα μελλοντικά μέτρα που θα περιλαμβάνει ο κανονισμός για τις επενδύσεις. Είναι κάτι από το οποίο έχουν να ωφεληθούν όλοι οι αλείς, οι ναυτικοί, είναι η ασφάλεια. Ακριβώς επειδή πρόκειται για μικρά σκάφη, ό,τι κάνουμε στον ε, μελλοντικό κανονισμό για την ενίσχυση της ασφάλειας εν πλώ είναι κάτι από το οποίο έχουν να υποφεληθούν όλοι, αλλά κυρίως η μικρή αλία. Τέλος για τη χρηματοδότηση, για τις οργανωτικές δραστηριότητες, για τις δραστηριότητες που επιτρέπουν στον τομέα να οργανωθεί καλύτερα, να οργανώσει τη διαχείρισή του, να βρει εναλλακτικέ και να οργανώσει συμπληρωματικές οικονομικές δραστηριότητες. Εδώ θα υπάρξει ένα μεγάλο εύρος ενισχύσεων που δεν αφορούν αποκλειστικά την μικρή αλία, αλλά θα υποφεληθεί ιδιαίτερα και η μικρή αλία. Αυτά. Και νομίζω τέλειωσε ο χρόνος μου, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, για 10 λεπτά, ο κύριος Μικέλο Τέγα από το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης. Αυτό θέλεις? Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, αξιότιμη προσκεκλημένη. Ονομάζομαι Μιγγέλ Λορτέγκα Σεδρά. Το πανεπιστημίου της Βαρκελόνης. Είμαι ερευνητής εκεί και θέλω να σας παρουσιάσω μερικές ιδέες για το πώς θα βελτιώσουμε την κοινωνικο-οικονομική βιωσιμότητα για να το επιτύχω αυτό θα προχωρήσω σε μια σύντομη εισαγωγή μετά σε ορισμένα οικονομικά στοιχεία και θα τελειώσω με συγκεκριμένε προτάσεις και συμπεράσματα. Η βασική ιδέα είναι η συνοχή. Η αλία μικρής κλίμακας μοιράζεται σε πολλές περιπτώσεις τους πόρους, τις αγορές, ε, την δημόσια χρηματοδότηση και τους κανονισμούς με τη βιομηχανική αλία. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε, διότι αυτός είναι ο βασικός στόχος ε, για τον οποίο δεν θα πρέπει να εφαρμόσουμε ε, επιπόλαια και με τμηματικά μέτρα, μερικά μέτρα τυχαία μέτρα δηλαδή στην αλία μικρής κλίμακας. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει συνοχή. Διαφορετικά δεν θα επιτύχουμε τους στόχους μας και δεν θα σεβαστούμε τους πολίτες μας. Για να επιτύχουμε όμως τη συνοχή πρέπει να ξέρουμε ακριβώς σε τι αρχές θα υιοθετήσουμε. Όπως είπαν προλαλήσαντες, όλοι συμμεριζόμαστε την ιδέα ότι αυτή η αλία μικρή κλίμακα αυτός ο στόλος, μπορεί, είναι ιδανικό για να αντιμετωπίσει την αλία η οποία έχει ελάχιστο, το ελάχιστο, τις ελάχιστες κακές επιπτώσεις στο περιβάλλον, η οποία μπορεί λίγα αποτελεσματικά να διανύμει την ευημερία και να σεβαστεί πολιτιστικά στοιχεία. Γι' αυτό λοιπόν αυτά τα στοιχεία, αυτές οι βασικές αρχές είναι πολύ σημαντικές ε, για την καλή αλία και τις καλές οικονομικές αποδόσεις. Για να επιτύχουμε λοιπόν την βέλτιστη αλλιευτική οικονομία πρέπει να παρουσιάσω ορισμένα κριτήρια, ορισμένα στοιχεία τα οποία είναι προϋπόθεση επιτυχίας. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι τιμές εξαρτώνται από την προσφορά και τη ζήτηση. Όμως υπάρχουν και πολλά άλλα στοιχεία που διαμορφώνουν την τιμολόγηση που μπορεί όμως να μην έχουν τελική, τελική επίπτωση στα αλλιέσματα. Η διαμόρφωση των τιμών εξαρτάται από τις ε, περιβαλλοντικές και κοινωνικές ε, εξωτερικές, ε, από τους εξωτερικούς παράγοντες. Για να είμαι πιο συγκεκριμένος, όταν μιλάμε για εξωτερικούς παράγοντες έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Το πρώτο είναι η διατήρηση μιας ισορροπίας, εδαφικής ισορροπίας και η ανάλυση της επίπτωσης ε, της αλίας στις κοινωνικο-οικονομικές δομές των παρακτήων κοινοτήτων. Ε, ε, ε, πρέπει λοιπόν αυτά τα δύο κριτήρια να τα λάβουμε υπόψη γιατί είναι εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση των τιμών. Επίσης σημαντικό είναι να, να γνωρίσουμε την, ποσοτικο, τη δυνατότητα ποσοτικοποίησης των εξωτερικών αυτών προϋποθέσεων. Είναι γεγονό ότι η αλία μικρής κλίμακος έχει τα πιο αποδοτικά σκάφη. και έχουν γίνει ε, μία πρόσθετη μελέτη έχει ακριβώς αξιολογήσει αυτές τις οικονομικές επιπτώσεις. Η βασική ιδέα είναι ότι δεν μπορούμε πλέον να γνωρούμε αυτές τις εξωτερικές επιρροές. Εάν θέλουμε να εφαρμόσουμε σωστά οικονομικά στοιχεία πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ε, αυτά, αυτοί οι εξωτερικοί παράγοντες υπάρχουν και ας εξετάσουμε γιατί λοιπόν είναι τόσο σημαντικά αυτά τα εξωτερικά στοιχεία. When do we have important externalities as Εφόσον λοιπόν αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες που έχουν σημαντικές επιπτώσεις, θα πρέπει να δεχτούμε ότι αυτές, αυτοί οι εξωτερικοί παράγοντες συνδέουν τα άτομα με, τις, ε, με την δημόσια πραγματικότητα. μόνο εάν υπάρχουν ωφέλη της, ε, από την αλληλεία τα οποία δεν οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες μπορούμε να δεχτούμε ότι δεν αγνοούμε τη μελέτη αυτών των παραγόντων. Αυτό όμως δεν γίνεται. Ε, οι, εξωτερικοί παράγοντες σίγουρα επηρεάζουν κάθε πτυχή της αλληλείας άρα πρέπει να τα θεωρήσουμε ως εξωτερικά μέσα, εξωτερικά εργαλεία. Σήμερα το πρωί ελέγχθη ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη τα, το ιστορικό υπόβεθρο, τα ιστορικά δικαιώματα και το παρελθόν αυτής της παράκτειας και αλίας μικρής κλίμακας. Αλλά εγώ πιστεύω ότι εκτός από τα ιστορικά, ε, ιστορικά στοιχεία πρέπει τώρα ο, περισσότερο από ποτέ να μελετήσουμε τους εξωτερικούς παράγοντες. Ε, χρειαζόμαστε εναλλακτικέ μεθόδους αλίας ε, και Γι' αυτό πρέπει να και συγκεκριμένα μέτρα. Για τα, αν εφαρμοστούν αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα θα εφαρμοστεί ένα δίκαιο επίπεδο δραστηριότητας, μια θεμητή αλληλεία δηλαδή, η οποία θα βασίζεται λιγότερο σε εξωτερικά στοιχεία. Πρέπει λοιπόν να μειώσουμε τα δυσμενή, τους δυσμενείς εξωτερικούς παράγοντες και να εισάγουμε στις μελέτες μας θετικούς εξωτερικούς παράγοντες όπως ενώσεις καταναλωτών, ενώσεις πολιτών, ε, άλλες συνεταιρισμού και ενώσεις. Πώς μπορούμε λοιπόν να το κάνουμε αυτό. Θα αναφέρω τρία θέματα. Η πρώτη ιδέα είναι ότι είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε θετικούς εξωτερικούς παράγοντες. Αλλά πρέπει να κάνουμε τη διανομή των πόρων, κατανομή των πόρων, συγγνώμη, με διαφορετικό τρόπο. Εάν δεχθούμε την εισαγωγή περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων, μπορούμε να μειώσουμε το ποσοστό των κακών εξωτερικών παραγόντων. Ορισμένα από τα κριτήρια που πρέπει να προσέξουμε αναφέρονται σε αυτή τη διαφάνεια. Τα βλέπετε. Πρέπει να εφαρμόσουμε μία αλία με χαμηλά επίπεδα περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με χαμηλά επίπεδα απορρίψεων, με χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακο, με καλή εφαρμογή ε, της νομοθεσίας, συμβατότητα και σεβασμό της νομοθεσίας και με ψηλό επίπεδο απασχόλησης. Η εισαγωγή περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων είναι ένας μηχανισ... συνεχής ε, μηχανισμός ε, ο οποίος θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με την εξέλιξη των εξωτερικών παραγόντων. Επίσης θα μπορεί να χρησιμεύσει σε, όλες τις... σε όλα τα είδη των στόλων και επίσης θα ε, ενισχύσει την παραγωγικότητα και τον ανταγωνισμό εντός και εκτός των αλληλευτικών στόλων. Τρίτον, ε, εισάγει τη συνοχή. Ακριβώς εδώ, αυτή είναι η ουσία όλου του θέματος, δεν είναι μόνο να δώσουμε χρήματα και οικονομικά μέσα, αλλά πρέπει να εφαρμόσουμε μία προοπτική συνοχής Πώς μπορούμε λοιπόν σωστά και συνεκτικά να εφαρμόσουμε αυτά τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Θα αναφέρω μερικούς τρόπους εισαγωγής. Δεν μας επαρκεί ο χρόνος να αναφέρω όλους τους τρόπους εφαρμογής, οπότε θα αναφέρω τους τρεις πιο σημαντικούς. Καταρχάς μπορούμε να κάνουμε την εισαγωγή αυτών των κριτηρίων στους βασικούς κανονισμούς ως γενικό κανόνα πολιετών προγραμμάτων. Βεβαίως τα πράγματα αλλάζουν από ένα πολιετές πρόγραμμα στο επόμενο. Αυτό είναι ένας καλός τρόπος αντιμετώπισης της ε, ποικιλομορφίας της αλίας αλλά όποια μορφή και αλίας, ε, ε, αν, ε, για όποια μορφή και να μιλάμε, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε την εισαγωγή αυτών των βασικών κριτηρίων. Επίσης πρέπει να εισάγουμε αυτά τα κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τις αληφτικές δυνατότητες και την κατανομή αληφτικών δυνατοτήτων. Μέχρι τώρα η Κομισιόν έχει προτείνει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να διατηρήσουν μέχρι ένα 5% ε, απόθεμα, το οποίο να αυξάνεται προοδευτικά. Ε, αυτό το ποσοστό λοιπόν μπορεί, επιτρέπεται να αυξηθεί προοδευτικά, αλλά μόνο εάν ληφθούν υπόψη τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Αυτό θα στείλει ένα σαφέστατο μήνυμα προς την σωστή κατεύθυνση. Και τρίτον, Πρέπει να διασυνδέσουμε τα χρηματοδοτικά μέσα με αυτά τα κριτήρια. Όσοι έχουν την καλύτερη απόδοση, το καλύτερο ιστορικό, ας πούμε, την πιο σωστή εφαρμογή των κριτήριων θα μπορούν να αποφεληθούν και από ε, την υπάρχουσα χρηματοδότηση. Με, μετά από αυτές τις τρεις συγκεκριμένε προτάσεις θα αναφερθώ πολύ σύντομα σε περισσότερες δράσεις ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Η αλία μικρής κλίμακος ε, μπορεί να αντέξει περισσότερα οικολογικά σοκ, οικολογικές αναμπουμπούλες. Η τρέχουσα πρόταση της Κομισιόν περιλαμβάνει ορισμένες ενδιαφέρουσες προτάσεις, αλλά περισσότερα πρέπει να γίνουν. Πρώτον, πρέπει σαφέστατα να υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα. Η αλία μικρής κλίμακος δεν μπορεί να περιμένει εσάι. Και αυτό είναι, αυτό υπάρχει και μία επιστημονική δικαιολόγηση. Ε, η αβεβαιότητα επιδεινώνει ένα περίπλοκο τομέα περαιτέρω. Δεύτερον, πρέπει να καθορίσουμε ποιες θα είναι οι ενδιάμεσες διαδικασίες μέχρι ότου ολοκληρωθούν οι τελικές προτάσεις. Το, το, το μεσοπρόθεσμο λοιπόν διάστημα πρέπει οπωσδήποτε να συνδεθεί με τα προαναφερθέντα κριτήρια. Τρίτον, αυτό το γενικό πρόγραμμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερεμένων πλευρών. Χρειαζόμαστε λοιπόν διαχειριστικές επιτροπές στο επίπεδο της αλίας. Ο, ο, διακόπτη η πρόεδρος, ναι, ξέρω, ξέρω, έχω ξεπεράσει το χρόνο μου. Ο τρίτος λοιπόν άξονας, η, η τρίτη δέσμη ενεργειών, είναι να, να συμπεριλάβουμε την, αρχή, την προληπτική αρχή και την, οικο, την, την προσέγγιση που βασίζεται στα οικοσυστήματα και στο σεβασμό της των αηφόρων συμφωνιών, αλίας. Γιατί λοιπόν τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια είναι απαραίτητα. Είναι απαραίτητα ε, διότι ε, παρουσιάζουν και οικονομικά πλεονεκτήματα. Ε, διευκολύνουν τη μείωση των κακών εξωτερικών παραγόντων και ωφελούν αυτούς που εφαρμόζουν τις καλύτερες πρακτικές. Δεν είναι θέμα μεγέθους, είναι η συμπερίληψη κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων ε, ε, ισότιμη με την εφαρμογή οικονομικών κριτηρίων. Ε, ξέρω ότι υπάρχουν πολλές άλλες προτάσεις στο τραπέζι μας και η πρόταση αυτή, το ψήφισμα αυτό που παρουσιάζει ο κύριος Ομπράιαν είναι εξαιρετικά καλό και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Φρεντερίκο Περέιρα τώρα έχει το λόγο που είναι πρόεδρος μιας οργάνωσης της Πορτογαλίας. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά ελπίζω. Γεια σας. Θα ήθελα να πω ότι δεν θα επιμείνω στο, στα χαρακτηριστικά της ε, μικρής της ε, παράκτης αλληλείας, αλλά είναι αλήθεια ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις ε, ευρωπαϊκές ε, περιφέρειες και ότι η αλληλεία επιτρέπει την επιδίωση των παράκτιων κοινοτήτων. Εμείς έχουμε πάνω από 9.000 ε, πλοιάρια, διαφορές ανάμεσα στις περιοχές με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στην Πορτογαλία η αλία, η παράκτη αυτή αλία ε, εκπροσωπεί 1% των πλοίων και 10% των ε, αλλιευμάτων. Και ε, τα πλοία τα οποία έχουν πολλαπλή δραστηριότητα θα λέγαμε, αποτελούν το 98% το, του στόλου και 40% των ε, ε, αλλιευμάτων. Τώρα, έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά που ανέφερα και το, τα οποία μας κάνουν να σκεφτούμε δεν μπορούμε να κάνουμε δεχτή την πρόταση της Επιτροπής. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι μικροί παραδοσία και παράλληλη αλληλεία είναι σημαντικές, αλλά τις θεωρεί μια άλλη κατηγορία και δεν υπάρχει σωστή υποστήριξη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φαίνεται να πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση, την ίδια. Θα πρέπει λοιπόν να αναθεωρήσει το ρόλο του, διότι ο ρόλος του είναι να υποστηρίξει του, τις μικρές κοινότητες. Θα πρέπει όντω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει με ζαφήνη από την Επιτροπή να αναγνωρίσει αυτή την ιδιαιτερότητα της παράκτεια και παραδοσιακής αλίας στην κοινή αλληλευτική πολιτική. Και επίσης η Επιτροπή να παρουσιάσει μια επιτροπή να παρουσιάσει Επιτροπή ένα ειδικό πρόγραμμα για αυτές τι δραστηριότητες για να αντιμετωπίσει, ε, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτού του τομέα. Κάτι το οποίο δεν βλέπουμε στην πρόταση αναθεώρησης που έχουμε από την Επιτροπή. Επίσης, το, ε, την επιφύλαξη για το θέμα των 12 ναυτικών μιλίων. Εμείς θεωρούμε θα πρέπει να επεκταθεί στα 24 για να μην πω 50 μίλια σε σχέση ό,τι ισχύει δηλαδή για τον κανονισμό για τις ε, απομακρυνμένες ε, και περιφερειακές περιοχές. Εμείς πάντοτε το λέγαμε όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων θα πρέπει να υπάρχει μια διαχείριση ε, αποκεντρωπημένη επιτόπου που λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας, κάθε ζώνης, κάθε στόλου και κυρίως να μπορέσουν να συμμετάσχουν ε, οι αλληλείς στη διαχείριση των πόρων. Αυτό θα πρέπει να υποστηριχθεί και ε, με επιστημονικό τρόπο. Θα πρέπει να γίνουν έρευνες, εργαστήρια να σκύψουν πάνω αυτό το θέμα, διότι χωρίς επιστημονική προσέγγιση δεν μπορεί να υπάρχει σωστή διαχείριση της αλίας. Επιπλέον, η συμμετοχή των αλλιέων σε αυτή τη διαχείριση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Κάτι το οποίο δεν βλέπουμε σήμερα. Ε, έκανα αναφορά σε ένα ψήφισμα ε, το οποίο επιμένει στην αναγκαιότητα ε, συμμετοχής των επαγγελματικών οργανισμών ε, ώστε οι αλληλείς να έχουν και αυτή την ευθύνη τους, να επομισούν ευθύνες. Το Κοινοβούλιο ζήτησε μεγαλύτερη, μεγαλύτερη αποκέντρωση, ούτω ώστε η, η εκπροσώπηση των αλληλείων να είναι σωστή. Διότι αυτοί εκπροσωπούν τις οπικές κοινότητες, ξέρετε. Να. Το να μειωθεί ο ρόλος, ο, συμβουλευτι... ο ρόλος των αλληλείων στι συμβουλευτικέ επιτροπές, κάτι το οποίο έχει γίνει μέχρι τώρα, είναι ειλικρινά κάτι το οποίο δεν, είναι, ε, δεν αρκεί, δεν είναι αποδεκτό. Στην πρόταση τώρα της Επιτροπής όσον αφορά τις ποσοστώσεις το γεγονός για την ιδιότητα δηλαδή που έχουν αυτές τις ποσοστώσεις να, είναι, ε, να μεταφέρονται. Έχουμε πολλά πλοία στη μικρή αλληλευτική δραστηριότητα και η Επιτροπή η ίδια είναι, έχει, είναι γνώστης ε, ότι με αυτή τις προτάσεις θα οδηγήσει σε, μια, σε ένα συγκεντρωτισμό όσον αφορά την αλία. Θα οδηγηθούμε σε μια ολιγαρχία θα έλεγα σε αυτό το τομέα της αλίας. Τώρα, για δύο άλλες πτυχές της ε, μεταρρύθμισης, οι οποίες δεν έχουν ίσως να κάνουν με την παράκτεια και μικρή ε, αλία, αλλά είναι σημαντικές για, αυτές, για αυτούς τους τομείς, παρόλα αυτά. Πρώτον, Μέχρι τώρα μας λέγανε ότι η κοινή αλληλευτική πολιτική είναι ένα σύνολο κανονισμών που έχουν να κάνουν με την διατήρηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη των πορών της αλίας. Για την οργάνωση της αγοράς της αλίας και σωστή χρηματοδότηση και διαχείριση. Σήμερα ο νέος κανονισμός όσον αφορά ε, τη χρηματοδότηση αντικαθιστεί το προηγούμενο. Και βλέπουμε ότι εδώ πέρα δεν γίνονται κάποιες ε, αλλαγέ. Θα θέλαμε να ξέρουμε αν αυτή η κοινή αλληλευτική πολιτική είναι συνώνυμη με τη βιώσιμη ανάπτυξη, ναι ή όχι. Ερώτημα πολύ ουσιαστικό. Για μας η διαχείριση των πόρων είναι βασική σημασία. Είναι απαραίτητη για την βιώσιμη ανάπτυξη, τη διατήρηση των πόρων και να εξασφαλίσουμε και το μέλλον τη Ελία. Αλλά είναι σαφέστατο ότι δεν μπορεί να είναι ο μόνος, ε, το μόνο θέμα το οποίο καθορίζει την πολιτική. Επίσης, η αλφτική πολιτική θα πρέπει να έχει σαν πρώτο στόχο, θα έχει να κάνει την, ε, ε την ε, προστασία φυσικά των πόρων, αλλά την προστασία των κοινοτήτων που ζουν από αυτήν την αλία. Ε, αυτά που βλέπουμε όμως οδηγούν προς την ε, αντίθετη κατεύθυνση και θα υπάρχουν επιπτώσεις ε, επιπτώσεις σε όλα τα άρθρα τα οποία θα ακολουθήσουν. Γι' αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να τοποποιηθεί αυτός ο κανονισμός όσον αφορά την μικρή αλεία. Γι' αυτό και θα τελειώσω θεωρούμε ότι αυτή η πρόταση κανονισμού ε, δεν λαμβάνει υπόψη όσον αφορά την, ε, τους ε, ιδιοκτήτες πλοίων, όπου για να γίνει διαχωρισμός όσον αφορά τη μικρή αλληλευτική δραστηριότητα. Να θα πρέπει να ληφθούν όλα τα στοιχεία τα οποία θα είναι σημαντικά. Ε, το θέμα το οποίο έχει να κάνει με, επίσης με τα καύσιμα που έχει και αυτό επιπτώσει στο κόστος. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Είναι σημαντικά για την βιωσιμότητα αυτού του τομέα. Κάτι το οποίο δεν γίνεται στη σημερινή πρόταση κανονισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο Χωσέ Λουίς Ροντρίγκες τώρα έχει το λόγο για 10 λεπτά από την Ισπανία. Παρακαλώ κύριε Ροντρίγκες, 10 λεπτά. Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Ονομάζομαι Χωσέ Λουί Ροδρίγες, είμαι μικρό αλίας από τη Γαλλικία της Ισπανίας και συμμετέχω στην σχετική οργάνωση της περιοχή μου. Είμαι από την Γαλλικία και αυτά που θα σας πω έχουν να κάνουν ως επιτοπλίστων με την περιοχή αυτή που γνωρίζω και καλά. Παρ' όλα αυτά, τα πράγματα θα μπορούσα να πω και για οποιαδήποτε άλλη παράκτια αλία της Ευρώπης. Στη Γαλλικία η μικρή κλίμακα σελία αποτελείται από διάφορους τομείς. Είμαστε πάνω από 4.000 ε, σκάφη, παραπάνω όπως βλέπετε. 12.000 ναυτικοί και οστρακοσυλλέκτες με παραπάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Είμαστε ένας δυναμικός, σύγχρονος τομέας με διαφοροποίηση της δραστηριότητές μας και εμπορία. Έχουμε πετύχει να τρέφουμε τίθυρα μαλάκια, κεφαλόποδα, οστρακοειδή. Μια άλλη δραστηριότητά μας βέβαια είναι τα κιδόνια πάρα Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι έχουμε κάνει την οικονομία μας ιδιαίτερα παραγωγική. Σε διάφορα σημεία της περιοχής μας δραστηριοποιούμαστε και πουλάμε απευθείας στον καταναλωτή πολλές φορές. Μάθαμε επίσης να διαφοροποιούμε την δραστηριότητά μας, συμπεριλαμβάνοντας τον τουρισμό, εκτός από την ε, αλία. Εμείς επεξεργαζόμαστε τα προϊόντα μας για να τα διαθέτουμε στην αγορά. Σας μίλησα για τον τουρισμό. Όντως δραστηριοποιούμαστε και στον τουρισμό. Πράγμα που σημαίνει ότι η δραστηριότητά μας αποκτά μεγαλύτερη αξία. Παρόλη την ε, μόλυνση των ποταμών και των ε, θαλασσών στα παράκτια της περιοχής μας, παρόλα αυτά έχουμε καταφέρει να διατηρήσουμε μεγάλη βιοποικιλότητα. Υπάρχουν οικότοποι στην περιοχή αυτή του πλανήτη μας και σε πάρα πολλές ζώνες μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε. Στην οργάνωσή μας για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την δραστηριότητά μας από το 2007 έχουμε ξεκινήσει με ένα πρόγραμμα που καθαρίζει τα ποτάμια και τις ακτές από κάθε είδους ρήπανση. Μας βοηθούν σε αυτό οικολογικές οργανώσεις, σχολεία, ώστε να βελτιωθεί το περιβάλλον και ώστε όλοι να μπορούμε να επωφεληθούμε και όχι να ζούμε μέσα σε ένα σκουπιδότοπο. Όπως ε, λοιπόν καταλαβαίνετε, τα χαρακτηριστικά της μικρής αλίας τη διακρίνουν από την αλία γενικά και μπορεί να αποτελέσει μια βιώσιμη δραστηριότητα. Δυστυχώς όμως αυτό δεν το έχει λάβει υπόψη της ε, η νέα κοινή πολιτική με μεθόδους που δεν ανταποκρίνονται σε αυτήν ειδικά. Πράγμα που δυσκολεύει πάρα πολύ τη ζωή μας. Οι πολιτικές που εφαρμόζονται δεν συνάδουν με τις ανάγκες της αλίας αυτής, ούτε με την προσφορά της, αλλά με άλλες αλίες οι οποίες δεν έχουν ούτε οικονομικό, ούτε οικονομικό, ούτε περιβαλλοντικό χαρακτήρα όπως έχει η μικρή αλία. Από το 2009 ξεκινήσαμε να δουλεύουμε για να ετοιμάσουμε ένα πρόχειρο για τη μεταρρύθμιση της κοινή ελευτικής πολιτικής. Με την πράσινη βίβλο εμείς τονίσαμε ποια είναι τα δικά μας τα κριτήρια. 2010 και 2011 γίνανε πολλές προτάσεις, συναντήσεις, πλατφόρμες για να προχωρήσει το σημείωμα μας αυτό. Συναντηθήκαμε με περιβαλλοντολόγους, οικολόγους, επιστημόνες κλπ. Και αυτό για να ενισχυθεί η μικρή αλία, ως βιώσιμη αλία που είναι. Και η νέα ΚΑΠ να τη χρησιμοποιήσει σαν μοντέλο. Τον Ιούλιο που μας πέρασε δημοσιοποίησαμε το πρώτο μας ε, πρόχειρο και διαπιστώσαμε ότι η ΚΑΠ δεν αναφέρει τίποτα γι' αυτό. Δυστυχώς μείναμε στους ευσεβείς πόθους και στις καλές προθέσεις. Γιατί στην πράξη δεν αναφέρεται αυτό το μοντέλο αλία στην ΕΑΚΑΠ. Οπότε να ρωτιόμαστε πώς τελικά θα ενισχυθεί η μικρή αλία εφόσον δεν αναφέρεται σχεδόν καθόλου στην ΕΑΚΑΠ, εφόσον δεν καθορίζονται κριτήρια, πώς θα υπάρξει διαφορετική μεταχείριση σε αυτήν εφόσον δεν διαφοροποιείται, δεν ορίζεται διαφορετικά. Υπάρχουν ε, κάποιοι παράγοντες οι οποίοι ήταν αποφασιστικοί γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα, η δυνατότητα που έχει ο τομέας να ενώνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρέπει, για να μπορούμε να πιέσουμε, να είμαστε ενωμένοι, ξεκινώντας από το Κοινοβούλιο. Έπειτα, μια άλλη διαπίστωση είναι ότι δεν υπάρχει μια πλατφόρμα διεκδικήσεων που να είναι ξεκάθαρη και που να καλύπτει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Αλία Μικρής Κλίμακας. Αν το κάνουμε χωριστά αναζώνει, χάνουμε σε δύναμη και θα χάσουμε τους στόχους μας. Δεν θα λυθούν υπόψη στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Πρέπει να προχωρήσουμε λοιπόν ενωμένοι. να έχουμε ένα ρεαλιστικό όραμα που λαμβάνει υπόψη το παρελθόν. Έχει συμμετάσχει σε πολλές συναντήσεις ο κλάδος. Το θέμα δεν είναι κάθε φορά να λέμε γιατί χάσαμε τις προηγούμενες φορές, αλλά να διαπιστώσουμε ότι μέχρι τώρα δεν καταφέραμε τίποτα. Ούτε με την προετοιμασία που κάναμε δεν καταφέραμε να πείσουμε ότι είμαστε ένας τομέας που πρέπει να τον ε, λαμβάνουμε υπόψη μας, παρόλο που το 80% του κοινοτικού στόλου είναι μικρής κλίμακας αλεία. Συνεπώς, από την οργάνωσή μας πιστεύουμε ότι επιγόντως πρέπει να οργανωθεί μια ευρωπαϊκή διάσκεψη για την μικρή κλίμακα αλεία, όπου να συμμετέχουν όλες οι ευρωπαϊκές οργανώσεις και να θέσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο τομέα, με προτάσεις πρωτοβουλίες και προγράμματα ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες αυτές και να διεκδικήσουμε την σωστή μεταχείριση από την Ευρώπη. Επήγει, συνεπώς, η δημιουργία μιας διεκδικητικής πλαταφόρμας όσον αφορά την μικρή αλία. Με συγκεκριμένο ορισμό πλήρη του τι είναι ευρωπαϊκή αλία μικρής κλίμακας. Δεν είναι σωστό να εφαρμόζουμε τις ίδιες προδιαγραφές σε όλους τους τόλους, χωρίς να γνωρίζουμε συγκεκριμένα τι ανάγκες έχουν οι... τα είδη αλίας που είναι πιο βιώσιμα. Άρα πρέπει να δημιουργηθούν διαφορετικά συστήματα διαχείρισης και ένα διαφορετικό ταμείο που να απευθύνεται στην μικρή αλία και να υπάρξουν κατάλογοι με ειδικά μέτρα για την ανάπτυξη της μικρής αυτής αλίας πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται σήμερα δεν έχουν συνεισφέρει μέχρι τώρα στην ανάπτυξη της μικρής αλίας, αλλά ενίσχυσαν τους μεγάλους στόλους, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό κάνουν υπερεκμετάλλευση. Να λάβουμε υπόψη μας το πού αλλιεύουν οι μεγάλοι αυτοί στόλοι και να λάβουμε υπόψη μας την απόσταση από ε, τα σημεία όπου αλλιεύουν οι μικροί στόλοι. Δεν πρέπει να υπάρχει αδράνεια πρέπει να στηρίξουμε την μικρή αλία. Δεν μπορεί να πληρώνουμε εμείς τη ζημιά που έχουν προκαλέσει άλλοι. Επιπλέον πρέπει να δημιουργηθούν συμμαχίες με παραφερείς τομείς, με τομείς που θέλουν την μικρή αλία. Τα δύο τελευταία χρόνια διαπιστώσαμε ότι πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις μιλούν υπέρ της μικρής αλίας και το κάνουν γιατί πιστεύουν ότι είναι μια βιώσιμη αλία, ότι έχει δυνατότητες ανάπτυξης. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε ότι μεταξύ μας πρέπει να υπάρχει συμμαχία, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας υπέρ της μικρής αλίας και έτσι οι επιστήμονες που παρακολουθούν την κατάσταση ε, θα πούν αυτό που λέμε και εμείς, ότι πρέπει να στηρίξουμε την μικρή αλία και να σχεδιάσουμε τον μέλλον μας βασιζόμενοι σε, στην αηφόρο ανάπτυξη και στην προστασία των πόρων. Εμείς πρέπει να κάνουμε τη φωνή μας να ακουστεί. Μέχρι τώρα δεν το καταφέραμε. Δεν καταφέραμε να περάσουμε τις απόψεις μας, τις ιδέες μας. Δεν ξέρω αν σήμερα μας ακούσατε. Η φωνή μας πρέπει να ενισχυθεί και να εμπλουτιστεί με επιχειρηματολογία, με απόψεις που θα κυκλοφορήσουν για να επιχειρηματολογούμε υπέρ της μικρής αλίας. Θέλουμε ένα μοντέλο μικρή αλίας σαν και αυτό που αναπτύσσουμε εμεί στην Γαλλικία. Για να μπορέσει όμω αυτό να μεταφερθεί οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη, πρέπει να πιστούν οι αλείς ότι έχει μέλλον το μοντέλο αυτό. Άρα είναι ευθύνη όλων η μελλοντική ΚΑΠ να χρησιμεύσει για τη διάδοση τέτοιων μορφών αλίας. Οι πολιτικοί, οι επιστήμονες, οι περιβαντολόγοι κλπ. κλπ. πρέπει να βοηθήσουν και όχι να αφήσουν το χρόνο να περνάει. Πρέπει να πετύχουμε το στόχο μας και αν μη τι άλλο να οριστεί μια ημερομηνία για να γίνει αυτή η διεθνής διάσκεψη που σας είπα για να ενισχυθεί η μικρή αλία. Ευχαριστώ. Yes. Ε, Ευχαριστούμε. Όλους τους ακούμε. Γι' αυτό είσαστε εδώ. Το Κοινοβούλιο τους ακούει όλους. Ακούει όλους τους κλάδους, όλους τους τομείς και εσάς. Τώρα, ο κύριος Ρωμέβα πρώτος που έχει στήσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ήθελα να πάρω το λόγο στο προηγούμενο πάνελ, προτίμησα να περιμένω μέχρι τώρα, αλλά έχω να πω τις εξής σκέψεις. Πρώτον, αυτό που ακούσαμε τώρα. Πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτή η ακρόαση που κάνουμε σήμερα. Πράγματι, από αυτό που ακούσαμε, όλοι καταλαβαίνουμε ότι το, κατά το παρελθόν το βάρος που είχε στις συζητήσεις η παράκτη αλία, η μικρή αλία, η παραδοσιακή, όπως ίσως καλύτερα πρέπει να ονομάζεται, ε, λοιπόν δεν είχε το βάρος το οποίο θα έπρεπε να έχει. Δεν την ακούσαμε αρκετά όσο θα έπρεπε. Καλό είναι λοιπόν που το κάνουμε αυτό σήμερα. Στα πλαίσια ε, προετοιμασίας της νομοθεσίας την οποία ετοιμάζουμε κι εμείς. Τώρα για τις ιδέες που άκουσα από τον κύριο Πένας για παράδειγμα όσον αφορά το Ταμείο. Όταν η Κομισιόν ξεκάθαρα λέει ότι θα είναι τα κράτη-μέλη τα οποία θα αποφασίζουν πώς, με ποιο τρόπο θα διαχειρίζονται τον τομέα και τους πόρους, εδώ υπάρχει μια παγίδα. Στην οποία κινδυνεύουμε να πέσουμε και εμείς και οι χώρες μέλη. Εντάξει, άμα πρέπει να το κάνουμε, να το κάνουμε. Ο κύριος Καντέκ δεν είναι τώρα εδώ, αλλά είπε ότι δεν πρέπει να βάζουμε σε αντιπαράθεση την ε, μεγάλη κλίμακα αλεία με την ε, άλλη μικρή κλίμακα. Εγώ νομίζω πως ναι, γιατί ο αντίκτυπος που έχει η μεγάλη αλεία σε σχέση με τη μικρή είναι τεράστιος. Άρα πρέπει να μειώσουμε κάποιες πρακτικές που επηρεάζουν το περιβάλλον για να προστατεύσουμε τα είδη. Άρα πρέπει να βοηθήσουμε τους μεν και να επιβάλλουμε κυρώσεις τους δε. Γι' αυτό χρειάζονται δύο πράγματα, τα οποία αναφέρθηκαν και τα επαναλαμβάνω ως προτάσεις που θα έπρεπε εμείς να προωθήσουμε με δικές μας τροπολογίες. Πρώτον, πολύ σωστά ζητάτε τη δημιουργία των επιτροπών συνδιαχείρισης, να είναι υποχρεωτικές. Ξέρω ότι έχουν περιορισμούς, δυσκολίες, αλλά αυτό που θέλουν οι μικροί στόλοι είναι οι αποφάσεις που λαμβάνονται να τυχαίνουν επεξεργασίες στο δικό τους επίπεδο, με επιτροπές διαχείρισης λοιπόν. Να υπάρχει φυσικά κάποια ευελιξία, γιατί πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας την πραγματικότητα επιτόπου, αλλά να μην περιοριζόμαστε στο σημερινό επίπεδο λήψη αποφάσεων, γιατί τότε αυτοί που θα μπορούν να επηρεάσουν περισσότερο θα είναι βέβαια οι πιο δυνατοί στόλοι, οι πιο μεγάλοι στόλοι. Η βιομηχανική αλία, μεγάλη κλίμακας λοιπόν. Συνεπώς, υποχρεωτικά αυτές οι επιτροπής ε, ε, συνδιαχείρισης. Έπειτα, κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι τα μακροπρόθεσμα σχέδια. Το είπε και ο κύριος Ορτέγκα τι κριτήρια θα υπερισχύσουν όταν αποφασίζουμε ποιος μπορεί να λιεύει πού. Αυτό έχει να κάνει με τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της δραστηριότητα και έχουμε χιλιάδες παραδείγματα και δεδομένα που δείχνουν ότι οικονομικά και κοινωνικά η μικρή αλία έχει πολύ θετικές επιπτώσεις. Αλλά και από πλευράς περιβάλλοντος καταστρέφει το περιβάλλον πολύ λιγότερο η μικρή αλία. Αυτά λοιπόν είναι κριτήρια τα οποία δεν μπορούν να μείνουν έτσι στον αέρα. Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα. Να τα συμπεριλάβουμε τα κριτήρια αυτά τα οποία θα καθορίζουν το ποιο τελικά έχει περισσότερο δικαίωμα στην αλία. Για να ποιος μπορεί να έχει μεγαλύτερη πρόσβαση στις ενισχύσεις, όπως έλεγε ο κύριος Πένας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ούτε εγώ πήρα το λόγο πριν στο προηγούμενο πάνελ, γιατί ήθελα να ακούσω όλες τις παρεμβάσεις. Όμως, σήμερα τι είδαμε. Είδαμε τι συμβαίνει στις διάφορες χώρες, στους διάφορους τομείς της Μικρής Αλίας. Και όπως είπε ο κύριος Πένα, Κοιτάξτε, πρέπει να αναγνωρίσω ότι εύκολα τα βάζουμε μαζί του, αλλά η μικρή αλία προστάθηκε τελευταία στιγμή στη μεταρρύθμιση. Οπότε εκείνος βέβαια είπε ότι παρόλο που της αφιερώνεται ένα μικρό κεφάλαιο δεν σημαίνει ότι δεν θα της αποδοθεί ένα διαφοροποιημένο καθεστώς διαχείρισης. Και μιλάει για τα 12 μέτρα σαν μοναδικό κριτήριο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξουν και άλλα, γιατί το κριτήριο δεν μπορεί να είναι μόνο ε, τα μέτρα του σκάφους, έχει να κάνει και με την ισχύ του κινητήρα του σκάφους, έχει να κάνει με τον εξοπλισμό που φέρει, έχει να κάνει με το πώς επηρεάζεται η τοπική κοινωνία οικονομικά και κοινωνικά από την αλία του εκάστοτε σκάφους. Τα κριτήρια είναι πολύ περισσότερα λοιπόν. Πώς θα θέσουμε σε εφαρμογή χωρίς κριτήρια ενισχύσεις. Θα είναι πολύ δύσκολο. Λέτε θα είναι ε, στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ε, όχι, αυτό είναι πολύ έτσι χαλαρό σαν και θα οδηγήσει σε διακρίσεις. Χάνουμε την ευκαιρία να έχουμε έναν ορθό ορισμό του τι είναι μικρής κλίμακας αλεία. Αυτό πρέπει να το θίξουμε. Μετά από αυτά που ακούσατε δεν μπορεί να μπαίνει σε ένα χωριστό έτσι μικρό κεφάλαιο η μικρή αλεία. Οι αλείς πρέπει να έχουν καλά προγράμματα διαχείρισης και γι' αυτό πρέπει να ληφθούν υπόψη περισσότερο και να τους δοθεί ένας συγκεκριμένο ορισμός που να τους διακρίνει βάσει και άλλων κριτηρίων, όχι μόνο των μέτρων των σκαφών. Ακούστε λοιπόν όσα είπαν ε, οι ομιλητές μας εδώ. Η κυρία Πατρονέβες τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε τόνισα ήδη πόσο σημαντικό είναι να διαφοροποιήσουμε μεταξύ της, να ξεχωρίσουμε την αλία μικρής κλίμακας από την αλία, ε, τη βιομηχανική ε, και ακριβώς η επιλογή κριτηρίων πρέπει να αποτελεί τη βάση ενός διαφοροποιημένου συστήματος. Υπήρχε παλιότερα στο θέμα αυτό μία ευρεία συνένεση στο Κοινοβούλιο ο κύριος Περέιρα είχε ε, αναφέρθηκε σε ένα έγγραφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2006. Το 2006 το Σώμα είχε ήδη τονίσει πόσο σημαντικό είναι να διαφοροποιήσουμε μεταξύ του, του αλλιευτικού στόλου και του, του βιομηχανικού στόλου και του, της αλλίας μικρής κλίμακος. Εμείς ε, είχαμε πει ότι μπορούμε κάτι να κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε μερικά πράγματα στην ε, με, μεταρρύθμιση αυτή της αλλιευτικής πολιτικής. Ζητήσαμε τη διαφοροποίηση μεταξύ αλλιευτικού στόλου, αλλιευτικής ε, βιομηχανικής αλλίας και αλλίας μικρής κλίμακας και η Κομισιόν δεν έκανε απολύτως τίποτα. Ε, τώρα είμαι ικανοποιημένη διότι παρατηρώ ότι η μικρή αλληλεία έχει τύχει μεγάλης προσοχής. Οπότε θέτω το ερώτημα πώς είναι δυνατόν αυτή η προϋπόθεση της θετικής διάκρισης να εφαρμοστεί στην αλία μικρής κλίμακας όταν δεν έχουμε ένα σαφή τι είναι βιομηχανική αλία και τι ακριβώς είναι η αλία μικρής κλίμακας. Πρέπει να βρούμε έναν ορισμό και να συμφωνήσουμε επ' αυτού. Ίσως το Συμβούλιο μπορεί να βοηθήσει. Υπάρχουν και μερικά κράτη-μέλη τα οποία δεν ενδιαφέρονται τόσο έντονα. Αλλά υπάρχουν άλλα κράτη-μέλη που πιστεύουν ότι αυτό το κριτήριο, αυτός, αυτός ο διαχωρισμός, η διαφοροποίηση μεταξύ δύο διαφορετικών τύπων αλίας πρέπει οπωσδήποτε να είναι σαφής, να οριστεί. Κατά την τελευταία μεταρρύθμιση Είχαμε συζητήσει την περιφερειοποίηση της κοινή ελευτικής πολιτικής. Πιστεύω ότι μπορούμε να αναδιαρθρώσουμε την περιφερειοποίηση αυτής της πολιτικής για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των διαφορετικών περιφερειών και ότι η κατάσταση είναι καλύτερα να κάνουμε μία αναδιάρθρωση της περιφερειοποίησης παρά να αφεύρουμε εντελώς νέα μέσα. Ε, ο στόχος μας είναι η απλούστευση και όχι η περαιτέρω περιπλοκότητα. Ευχαριστώ όλους τους ε, ομιλητές που μίλησαν σήμερα για τη βοήθειά τους, για την ενημέρωσή τους, για την παρουσίαση τόσων πολλών στοιχείων και ε, πιστεύω ότι μας έδωσαν το ένευσμα περαιτέρω εμβάσινση σε αυτό το τομέα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σαφώς ενήμερο ε, για τη σημασία της αλίας και τη σημασία των ε, εξελίξεων στον τομέα της αλίας και πρέπει να μας έχετε εμπιστοσύνη ότι θα κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της αλίας. Ο κύριος Φερέιρα. Ευχαριστώ. κυρία Πρόεδρε θεωρώ ότι αυτά που ακούσαμε ήταν πολύ σημαντικά και μας βοηθάει για να καταλάβουμε καλά την κατάσταση. Αν δεν, θέλετε, αν δεν θέλουν ατομικά δικαιώματα μεταφέρσιμα, μας μας πούνε στα ίσα και τι ακριβώς μπορεί να προβλέψει κανείς. Μια αναλλακτική λύση. Δεν μπορεί κανείς να μας πει ότι δεν υπάρχουν άλλες λύσεις. Μας εμπλούτησε αυτή η συζήτηση σήμερα και μπορούμε να έχουμε μια συζήτηση να δούμε εναλλακτικές λύσεις, να δούμε τα κοινωνικά δικαιώματα και να μπορέσει η παράκτια αλληλεία να πάει παραπέρα. Ε, θα πρέπει να γίνει μια διαβούλευση Απ' τη μια υπάρχει το θέμα της υπερβολικής ε, συγκέντρωσης. Δεν μας, λέει ακριβώς, δεν μας λένε τι ακριβώς θα γίνει και πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το ενδεχόμενο ρίσκο. Ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Σίγουρα θα πρέπει να δούμε τη δυνατότητα να έχουμε ε, μια δραστηριότητα η οποία είναι πιο βιώσιμη. Θα πρέπει να ξέρουμε δηλαδή τι ισχύει στον χώρο αυτό. Το αν μπορώ εγώ να ε, αλλιεύσω ή όχι ή κάποιος άλλος αν μπορεί να κάνει εις τη δική του δραστηριότητα. Υπάρχει κάποια ε, ζημία ίσως ε, όσον αφορά τα δικαιώματα να είναι μεταμέρσιμα, αλλά σίγουρα υπάρχουν και άλλες αναλλακτικές λύσεις. είναι σαφέστατο ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν αποκλείει όλα όσα έχουν να κάνουν με την παραδοσιακή αλία. Έχουν γίνει παρεμβάσεις και μέθοδοι έχουν... Έχει γίνει κατανοητό, υπάρχουν ε, κριτήρια, πράγματα που επιτρέπουν να έχουμε μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική δραστηριότητα. Επιτρέψτε μου και μια τελευταία ερώτηση. Αν... Σε σχέση με προλαλήσαντες, ε, πολλοί ομιλητές αναφερθήκανε αναφερθήκανε πολύ στο θέμα, ε, στο θέμα του εισοδήματος έγινε αναφορά ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα σε αυτή την παραδοσιακή αλία. Και εδώ πέρα η κοινή πολιτική θα πρέπει να παίξει ένα ουσιαστικό ρόλο. Ο κύριος Σίβενσον Φερρυπίν είπε ότι πώς θα προβληματιστούμε πάνω σε αυτό το θέμα, να εγγυηθούμε το ώστε ο καταναλωτής να, ε, να ανταμείψει αυτό το χαρακτήρα της βιώσιμη παραδοσιακής αλληλεία. Ε, υπάρχει αγορά. Η αγορά δεν ε, δίνει λύσει. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντε εξωτερικοί που επηρεάζουν τα πράγματα. Είμαστε σε μερίδιο κρίσης και ξέρουμε ότι ο, ο φτωχός καταναλωτής έχει τη... δεν ξέρει ε, κανείς αν έχει τις δυνατότητες να μπορέσει να ανταμείσει μια τέτοια δραστηριότητα. Ίσως θα πρέπει να γίνει της ε, ε, σαφής παρουσίαση ενδείξεις σε όσον αφορά αυτά τα προϊόντα. Θα πρέπει σίγουρα να, δούμε, να βρούμε κάποιους μεκανισμούς για να εξασφαλιστεί ένα μήνυμα, ένα ελάχιστο εισόδημα. Ευχαριστώ. Ο κύριος σας Ευχαριστώ η παραδοσιακή παράκτια αλία είναι αυτή που έχει περισσότερες κοινωνικές επιπτώσεις με περισσότερα σκάφη και είναι αυτή η οποία δραστηριοποιείται περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε κοινωτικό επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν όταν μιλάμε για τα 12 μέτρα για τις αλληλευτικές δραστηριότητες πρώτον επιβεβαιώνω ότι οι δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την συλλογή οστράκων θα συμπεριληφθούν. Η καλλιέργειά τους, γιατί και αυτοί έχουν οικονομικές επιπτώσεις. Δεύτερον, νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε κριτήρια επιλεξιμότητας στο τομέα αυτό της μικρής αλίας. Και τρίτον, να υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που να περιλαμβάνει και άλλα κριτήρια, όπως για παράδειγμα την ποιότητα των υδάτων. Πού είναι στοιχείο της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Η συλλογή οστράκων επηρέαζεται πάρα πολύ από την ποιότητα των ε, υδάτων. Και σε πολλές περιπτώσεις έχουμε δει τι προβλήματα έχουν ε, δημιουργηθεί. Ο κύριος Γκάλαγκερ. κυρία Πρόεδρε, είμαστε υποχρονική πίεση. Γι' αυτό, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή ήταν μια ευρεία συζήτηση και το, το πρωί ακούσαμε από την Κομισιόν. Αλλά όλη η μέρα σήμερα, πρωί και απόγευμα, ήταν μια πάρα πολύ καλή μέρα για την Αλία. Κάναμε μια εμπεριστατωμένη και εις συζήτηση για τη σημασία τις αλίες, τις παράκτιες περιοχές και στα, στις νησιώτικες περιοχές uh, και έχει μεταφέρει το βάρος από τη θεωρία στην πράξη. Το πρώτο πάνελ ε, ήταν πολύ επικοδομητικό, πολύ ε, ε, ενδιαφέρον και η συζήτηση που ακολούθησε και όλοι οι ομιλητές και στο επόμενο πάνελ ε, αναγνώρισαν τη σημασία της αλλίας μικρής κλίμακας. Είναι πολύ σημαντική να γίνεται αυτή η συζήτηση στην Επιτροπή Αλίας, διότι πρέπει εμείς τώρα να επιμείνουμε η παράκτη αλία και η αλία μικρής κλίμακας να συμπεριληφθεί στις προτάσεις της Κομισιόν και να σταματήσει ε, η η άρνηση της Κομισιόν και οι, οι, υποσχέσει υποσχέσεις της ότι θα τη συμπεριλάβει. Ε, είναι γεγονός ότι είναι μία, ένας ωφέλιμος τομέας αυτός που δημιουργεί θέσεις απασχόλησης και που μπορεί να αντιμετωπίσει σωστά το θέμα της εκμετάλλευσης πόρων που συνεχώς μειώνονται. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε την ευκαιρία σε αυτή την παράκτια και μικρή αλληλεία να χρησιμοποιήσει τους καλύτερους τρόπους για την, αηφόρο, για την επιβίωση βιωσιμότητα και αηφόρο ανάπτυξη της αλίας. ακούσαμε λοιπόν πάρα πολλά σωστά πράγματα σαν θα απαντήσουμε στην Κομισιόν και από αυτού θα κριθούμε. Θα κριθούμε για το ενδιαφέρον μας ε, για την Αλία. Ευχαριστούμε κύριε Καλεγέρ. Τώρα θα δώσω και πάλι το λόγο σε όσου ε, έκαναν τις παρουσιάσεις τους για να σχολιάσουν τα όσα ακούσαμε. Ο κύριος Πένες πρώτα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και για μένα ήταν μεγάλη χαρά που μπόρεσα να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση. Θέλω να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις που άκουσα. Πρώτον, πάνω από ένας αναφερθήκατε στα κριτήρια ε, κατανομής μέσα ε, στα κράτη-μέλη. Λες και η ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει το ζήτημα να το αφήσει στα κράτη-μέλη. Όχι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευχαρίστω να το ρυθμίζει αυτό σε κοινοτικό επίπεδο. Όμω υπάρχει μια μακρά παράδοση μέχρι τώρα που λέει ότι η εσωτερική κατανομή των δικαιωμάτων των εθνικών ποσοστώσεων γίνεται βάσει των κριτηρίων που καθορίζουν τα κράτη-μέλη. Μέσα στο κάθε κράτος μέλος. Αυτή είναι η παράδοση. Παρόλο λοιπόν που η ιδέα σας είναι ευπρόσδεκτη, σας διαβεβαιώ ότι στο Συμβούλιο των Υπουργών θα αποτύχει. Με τίποτα δεν πρόκειται να δεχτούν κάτι τέτοιο οι Υπουργοί. Να το ξέρετε. Σημειώνουμε επίσης και την ιδέα για την συνδιαχείριση. Τα σχέδια συνδιαχείρισης μπορεί να είναι μια λύση. Και το επαναλαμβάνω, το έχω ξαναπεί κυρία Πρόεδρε, ότι ένα από τα πράγματα που θέλουμε να πετύχουμε στα πλαίσια αυτής της ε, περιφερειακής διάστασης είναι να βρούμε μηχανισμούς συνδιαχείρισης που δεν είναι δυνατόν να τους έχουμε εδώ στις Βρυξέλλες. Σημειώνω επίσης και την ιδέα της κυρίας Πατρονέβες που λέει ότι δεν πρέπει να πολλαπλασιαστούν οι οργανισμοί και πρέπει να απλοποιήσουμε την πολιτική. Όταν συζητάμε, να συζητάμε, όταν συνεχίσουμε να συζητάμε με τα κράτη-μέλη για τις αποφάσεις όλων εκείνων των στοιχείων που έχουν να κάνουν ε, με την περιφερειακή διάσταση, αυτή είναι μια συζήτηση που δεν μπορεί ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να την καθορίσει συγκεκριμένα, γιατί τα κράτη-μέλη θα γυρίσουν και θα μας πούνε «Α, οι Βρυξέλλες ανακατεύονται στις αρμοδιότητές μας». Δεν θέλουμε να εμπλεχτούμε σε κάτι τέτοιο. Στο βαθμό πάντως που οι επιτροπές αυτές συνδιαχείρισης είναι αναγκαίες και τις θέλουν τα κράτη-μέλη, για την περιφερειακή συνεργασία, κανένα πρόβλημα. Και επιπλέον, σημαντικό αυτό, στην πρόταση του μελλοντικού δημοσιονομικού κανονισμού, μια από τις ιδέες είναι η δυνατότητα βοήθειας ώστε οι επαγγελματίες να μπορούν να συμμετέχουν στις, συνεδριώτες, στις συνεδριάσεις εκείνες όπου χρειάζεται να υπάρχει τοπικά μια διαχείριση. Δεν έχουμε πρόβλημα με αυτό. Αυτό όμως που δεν μπορώ να σας πω ότι πρέπει να νομοθετούμε από τις Βρυξέλλες. Όχι, εμείς θέλουμε απλοποίηση. Όλες οι ιδέες σας είναι ευπρόσδεκτες. Δεν σημαίνει ότι όλες θα συμπεριληφθούν σε ένα βασικό κανονισμό. Πολλές μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή πιο αποκεντρωμένα. Θέλω επίσης να αναφερθώ και σε κάτι άλλο που είπε ο κύριος Φερέιρα μετά. Είναι το κριτήριο των 12 μέτρων. Αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε κυρία Πρόεδρε. Γιατί μια που υπάρχουν πολλές πτυχές στην πρόταση αυτή που είναι θέματα αρχής για την Κομισιόν, η βιώσιμη δραστηριότητα, η δυνατότητα απορρίψου κλπ. Αυτά είναι θέματα αρχής για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά υπάρχουν και άλλα που έχουν να κάνουν με τα μέσα που χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, ποιο είναι το κριτήριο για να διακρίνουμε την μικρή αλία από την μη μικρή αλία. Θα μπορούσαν να υπάρχουν εκατοντάδες κριτήρια. Κανένα δεν θα ήταν τέλειο. Ούτε αυτό των 12 μέτρων είναι τέλειο. Αλλά και τα άλλα που εξετάσαμε ούτε και αυτά μας φάνηκαν τέλεια. Πρέπει όμως να υπάρχει ένα κριτήριο για να ε, διακρίνουμε τις δραστηριότητες και που να ε, επηρεάζουν τα μέτρα. Το κριτήριο αυτό πρέπει να είναι εύκολο, εφαρμόσιμο, για να ξέρουμε κατά πόσο συμμετέχει στο σύστημα το ποσοστό που μεταφέρονται ή όχι, αν πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, την ώρα, πόση ώρα κρατάει παλήρια, πόσο δεν ξέρω τι, καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι περίπλοκα κριτήρια και τότε η διαχείριση θα γινόταν πολύ πιο περίπλοκη, πιο δύσκολο ελεγχόμενη και όχι σταθερή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν δεν βάζει θέμα αρχή εδώ. Απλώ λέει ότι χρειαζόμαστε ένα απλό κριτήριο, σαφέ, για να διακρίνουμε τη μία δραστηριότητα από την άλλη. Κύριε Πρόεδρε, χρειάζεται αυτή η διαφοροποίηση, γι' αυτό. Αν υπάρχουν καλύτερες ιδέες, ευχαρίστω δεν είναι προκαταλημένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε έχει καμιά μόνη ιδέα να ενισώνει και καλά τα 12 μέτρα το κριτήριο. Απλώ θεωρεί ότι είναι ένα απλό κριτήριο και εύκολο εφαρμόσιμο. Αυτά κυρία Πρόεδρε. Τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε κύριε Σφαίρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο κύριος Ορτέγα, που μου δώσατε τη δυνατότητα να συμμετάσχω εδώ. Θέλω να αναφερθώ σε κάποιες στοιχείες που ακούστηκαν. Πρώτα απ' όλα δυσκολία καθορισμού κριτηρίου για τον ορισμό της μικρής αλίας. Είναι ένα θέμα που μας παιδεύει εδώ και πολύ καιρό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε το επιχείρημά μας που λέει ότι πρέπει να υπάρχει συνοχή στην ε, αλία μας. Να λαμβάνουμε υπόψη μας ε, τα πλεονεκτήματα της μικρής αλίας. Ξέρουμε ότι η διαφοροποίηση στις δραστηριότητες έχει σαν αποτέλεσμα ότι δεν θα μπορέσουν να καλυφθούν οι επιθυμίες του τομέα της μικρής αλίας. Αυτό τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Περέιρα τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν μου τέθηκαν συγκεκριμένα ερωτήματα, όμως ε, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τους διοργανωτές αυτής της συζήτησης και σας διαβεβαιώ ότι θα μεταφέρω την πεποίθησή σας στους αρμόδιους ότι η βιώσιμη αλληλεία ε, θα υποστηριχθεί από το σώμα και ότι το αξίζει, αξίζει την υποστήριξή σας. Αυτή είναι η πρώτη γενική παρατήρηση. Η αλληλεία μικρής κλίμακος είναι απόλυτα σχετική και ε, είναι, είναι πολύτιμη και πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθεί από τους ε, ε, κανονισμούς, από τους αντίστοιχους κανονισμούς. Και τέλος, ορισμένα, ορισμένες πτυχές που θεωρώ εγώ ιδιαίτερα σημαντικές. Πρώτον, πρέπει να δεχτούμε ότι η αλία μικρής κλίμακας ε, από ε, οικολογικής πλευρά προσφέρει εγγυήσεις βιωσιμότητας. Σέβεται ε, την τοπική πραγματικότητα, την, τους πόρους, τη σωστή διαχείριση των πόρων και τέλος το θέμα του, των εισοδημάτων, της διαφύλαξης των εισοδημάτων. Αυτό απασχολεί γενικά την αλία. Το εισόδημα των ε, ε, αλλιέων των, αυτών που συμμετέχουν στον τομέα ε, πρέπει να είναι βιώσιμο. Όλα τα μέτρα δεν θα πρέπει να φωλήσουν την, την γενικώ, αλλά και να ενισχύσουν το εισόδημα των εργαζομένων. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Κύριε Ροντρίγκε, η σειρά σας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ που μας προσκαλέσατε για να συμμετάσχουμε στη διάσκεψη αυτή. Μετά από αυτά που είπε και ο κύριος Ερνέστο Πένας Λάδο, θα ήταν σφάλμα εάν καθορίζαμε την μικρή αλία, λαμβάνοντας υπόψη μας ως κριτήριο μόνο το μήκος του σκάφους. Είναι λάθος. Πρέπει να αλλάξει αυτό να βάλουμε δύο, τρία, πέντε κριτήρια, πάντως όχι μόνο ένα κριτήριο, για να μπορέσουμε να διαφοροποιήσουμε μία αλία βιώσιμη, μία αλία χωρίς απορρίψεις. Και μέσα στο, στα σκάφη αυτά υπάρχουν και σκάφη με 9 μέτρα, αλλά και άλλα με 14 μέτρα. Αυτό λοιπόν λέμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να αλλάξει αυτό το σημείο και να ληφθούν υπόψη και άλλα κριτήρια τα κριτήρια που χρειάζονται για να ορίσουμε μια για πάντα την αλία μικρής κλίμακας. Αυτό το ζητάει ο κλάδος γιατί θέλουμε να ξέρουμε ποιες θα είναι οι πολιτικές που θα εφαρμοστούν, που θα έχουν οικονομικές επιπτώσεις, αλλά και αποφάσεις που θα έχουν να κάνουν με τις ποσοστώσεις. Πρόεδρος. Καλώς. Πέντε λεφτά έχω στη θέση μου για τα συμπεράσματα. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ όλους που συμμετείχατε στην ακρόαση αυτή. Νομίζω ότι ακούσαμε εδώ πολλές ιδέες. Φαντάζομαι οι συγητές για τα διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με τη μεταρρύθμιση θα τις λάβουν υπόψη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας βοηθήσατε με τη συζήτηση αυτή και έτσι Επιτροπή και Κοινοβούλιο ε, αντιλαμβάνονται τις θέσεις σας. Τώρα, συμπεράσματα είναι δύσκολο να καταλήξω σε συμπεράσματα, μια που ακούσαμε πολλές και διάφορες απόψεις. Αλλά το βέβαιο είναι ότι θα λάβουμε υπόψη μας τις παρατηρήσεις σας στις εργασίες μας. Τώρα, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Σε δύο-τρία πρέπει να τελειώσουμε. Οπότε περνάω στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξης, που είναι τα διάφορα. Δεν έχουμε. Σημείο 9. Ανακοινώσει της Προέδρου για τις αποφάσεις που πήραν οι συντονιστές χτε. Σας έχουν μοιραστεί οι προτάσεις. Κύριε Γκάλαγκερ, έχετε κάτι να πείτε σχετικά. Παρακαλώ κύριε Γκάλαγκερ. Και εγώ θέλω να επαναλάβω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή ημερίδα αυτή. Αλλά θέλω να σχολιάσω το σημείο 112 2-1-2. Α, το σημείο 1-1-2-2 που λέει ότι μπορούμε να αναθέσουμε, α, πώς, μπορούμε, πώς το αναθέτουμε τις γνωμοδοτήσεις. Τουλάχιστον ένας βαθμός ε, όταν κάποιος επιδείξει ενδιαφέρον. Εν πάση περιπτώσει, ε, μισός βαθμός για τη Γρυλανδία, ε, η ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών ζήτησε ένα από τα μέλη της να είναι εισηγητής αυτής της γνωμοδότησης. Δεν πρέπει κάποιος να θεωρήσει τις αποφάσεις των συντονιστών ως, δεδομένων, ως δεδομένες εφόσον δεν έχουν την τελική σφραγίδα από εμά. Είναι ένα διαδικαστικό θέμα και ζητώ τη συμβουλή, τη σας. Είναι μια νέα διαδικασία ή όχι. Αν δεν είναι καινούργια, τότε θα, θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θα δώσουμε ένα βαθμό ή μισό βαθμό σε αυτόν που είναι επόμενος στον κατάλογο. Eh, Συγγνώμη, η πρότασή σας τελικά συγκεκριμένα ποια είναι. Ένα πόντο να δώσετε, αυτό θέλετε να πείτε. Μα εγώ έλειπα. Οι συντονιστές και η Επιτροπή αποφάσισαν να αλλάξουν την πολιτική και να δίνουμε μισό πόντο. Εγώ νόμιζα ότι πάντα ήταν ολόκληρη πόντοι Ένας, δύο, τρεις. Μισό πόντο ή μηδέν πόντο ποτέ δεν είχαμε. Μετά περνούσαμε στο σύστημα εκπεριτροπής. Eh, η κυρία Πατρανέβες. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ο συντονιστής του ΕΛΚ, ο κύριος Ατινόρ, δεν ήταν παρόν. Και αυτό επέστησε την προσοχή μου σε αυτό. Χτες, στη συνεδρίαση των συντονιστών, ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση προσπάθησε να παρέμβει. Το κριτήριο για την κατανομή των εκθέσεων να πρέπει να ξεκινάει από το μισό της αξίας της έκθεσης, αλλά όχι πιο κάτω. Αν λοιπόν οι εκθέσεις που κατανέμονται, μοιράζονται και που αρχικά έχουν αξία δύο πόντους, τότε θα πρέπει να ε, γίνεται πλειοδότηση για ένα πόντο. Και αν ας πούμε για την Γουινέα Μπισάο που αξιολογήθηκε για δύο πόντους υπήρχαν δύο ομάδες που τη θέλανε. Με δύο πόντους ξεκινήσαμε για αυτή την έκθεση, αλλά τελικά καταλήξαμε να πληρώσουμε ένα πόντο, το μισό δηλαδή από την αρχική της αξία. Γι' αυτό και εγώ Σα έδωσα το παράδειγμα της Γουινέα Μπισάου γιατί ήταν μια έκθεση που αρχικά άξιζε δύο πόντου και κατέληξε ένα πόντο. Για τη Γρυλανδία είναι λιγότερο από το μισό της αξίας της που τελικά δόθηκε. Και αυτό δεν συνάδει με τον κανονισμό. Τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που λέει ο κύριος Γκάλεκερ. Πρόεδρος, Γουινέα Μπισάου είναι ένα πόντο, δεν είναι δύο πόντοι ένα πόντο και δόθηκε για ένα πόντο. Οπότε δεν είναι σωστό αυτό που λέτε εσείς. Δεύτερον, χτες για μισό πόντο δόθηκε η αλέκθεση και υπήρχε συνένεση. Δεν φταίω εγώ. Συμφώνησαν όλοι. Είπα χθε ό,τι είχα να πω, πάντω υπήρξε συμφωνία. Εσεί το αμφισβητείτε, εσεί το αμφισβητείτε. Υπάρχει και κανένα άλλο που αμφισβητεί το ότι δόθηκε οι σοσιαλιστέ για μισό πόντο. Γιατί τότε να ψηφίσουν οι παρόντες. Κύριε Λέβιν, τι έχετε να πείτε. Ευχαριστώ. Αυτό το πρόβλημα, ενημερώθηκα για αυτό το πρόβλημα μόλις τώρα και δεν ξέρω 100% σίγουρο τι λέει ο κανονισμός, αλλά βέβαια ε, εμείς θέλουμε να εφαρμοστεί ο κανονισμός. Εάν ο κανονισμός είναι ότι θα πέφτεις από, τα, τους δύο πόντους στον ένα και από το ένα στο, στο μηδέν, εντάξει, έστω. πολλά προβλήματα έχουν προσιαστεί με αυτό το θέμα, οπότε ας στηρίσουμε τους κανόνες, τον κανονισμό. Κύριε Στίβενσον, πρέπει να τελειώσουμε. Γρήγορα, παρακαλώ. Αυτό που θέλω να αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν υπάρχει προηγούμενο και αν έχουμε δώσει γνωμοδότηση για μισό βαθμό. Πόντο, συγγνώμη. Ένα πράγμα έχω εγώ να πω. Υπάρχουν κάποιοι κανόνε του παιχνιδιού που δεν τηρούνται. Γι' αυτό αποφασίζουμε με συνένεση. Γι' αυτό σα επαναλαμβάνω. Ό,τι θέλετε να τηρήσω από του κανόνε, αλλά υπήρξε συνένεση. Ενώ τώρα έρχεστε και το αμφισβητείτε. Ενώ χτε υπήρχε συμφωνία. Εγώ τι θέλετε να κάνω, να το ξαναψηφίσουμε άμα θέλετε αυτή την πρόταση. Αυτό έχω να πω. Παρακαλώ κύριε Μπρότσο. Έχετε το λόγο, αλλά πρέπει να τελειώσουμε γιατί οι διερμηνεί πληρώνονται για να δουλεύουν μέχρι τι 6.30, λέει ο Πρόεδρος. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ και για την υποστήριξή σου υποστήριξή σας. Εχθές κάνουμε μια έντονη συζήτηση ε, και, και, μου φαίνεται περίεργα αυτά τα οποία γίνονται τώρα. Και σημείωσα ότι καμία ομάδα δεν είχε ενδιαφέρον για αυτή την έκθεση και είπαμε ωραία θα πληρώσουμε μισό πόντο και θα το κάνουμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που για μισό πόντο παίρνουμε μία έκθεση ε, και δεν καταλαβαίνω γιατί ε, όλοι συμπεριφέρονται σαν να είναι αυτό κάτι εντελώς καινούριο. Ε, συμφωνήσαμε, αν όλοι είναι ευχαριστημένοι μπορούμε να δώσουμε άλλο μισό πόντο και να γίνει ένας πόντος, αλλά χτες δεν σημειώσαμε το ενδιαφέρον κανενός. Η πρόταση της κυρίας Πρώτος να δώσουμε σε ένα πόντο τη Γρυλανδία, νομίζω είναι κάτι που οικονοποιεί όλους τους παρόντες. Έτσι δεν είναι. Ωραία. Αυτό αποφασίζουμε λοιπόν και με αυτή την τροποποίηση εκεί μένει το πράγμα. Επόμενη συνεδρίαση 22 Νοεμβρίου εδώ στις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την παρουσία σας. Έληξε συνεδρίαση.